Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στην απογευματινή μου συνεδρίαση και χαίρομαι διότι έχουμε εδώ σήμερα τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης ε, ε, Ερεύνης, τον κύριο Ρόμπερτ Γιάν Σμίτς. Ελπίζω το πρόφερα σωστά. Ε, χαίρομαι για τη συνεργασία. Θα του δώσω τον χρόνο να κάνει την παρουσίασή του και μετά θα μπορέσουμε να συζητήσουμε ίσως κάποια θέματα. Ευχαριστώ κύριε Ρόιλ. Αγαπητοί ε, κύριοι, κυρίες και κύριοι, ε, χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα σαν νέος Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης ε, Ερεύνης και Καινοτομίας, γιατί από αύριο θα προσθεθεί και όρος καινοτομίας ε, είχατε μία επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Γκίγκαν Κουίν και είμαστε ε, όλοι ε, δεσμευμένοι να προωθήσουμε και να διαμορφώσουμε την πολιτική της Ευρώπης σε αυτούς τους τομείς. Δεν είμαι νεοφερμένος ούτε στην Επιτροπή, ούτε ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε σε αυτήν εδώ την Επιτροπή την Ήτρε και είχα ήδη πολλές επαφές με πολλούς από εσά, π.χ. με την κυρία Λοκατέλη για της, ε, ε, για, το πρόγραμμα πλαίσιο 7 με την ε, κυρία Μαντουρές, με την κυρία Νίμπλερ, με τον κύριο Βανίστελ Ρόις για τις διασυνδέσεις με το πρόγραμμα πλαίσιο και έτσι μπορώ να πω ότι είχα πολλές επαφές μαζί σας τα τελευταία χρόνια και πάντοτε είχαμε άμεσες επικοδομητικές παρόλο που δεν συμφωνούσαμε πάντοτε μπορούσαμε πάντοτε να προχωρήσουμε σε ένα πνεύμα διαλόγου. Θα ήθελα να σας πω πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή προετοιμάζοντας το πρόγραμμα πλαίσιο υπαριθμών 8 και ε, στο τέλος θα πω και μερικά λόγια σχετικά με το ίτερ που είναι το αγαπημένο μας θέμα διότι από όταν ε, με ε, διόρισαν κάθε μέρα έχω στο γραφείο μου το ίτερ τροπολογίες, προτάσεις, άρα είναι ένα πολύ φλέγον θέμα. Θα ήθελα εδώ όμως να συζητήσουμε το πρόγραμμα πλαίσιο 8 διότι αρχίζουμε κάνουμε τις πρώτες σκέψεις επί του θέματος αυτού και μας απασχολεί η ε, διαμόρφωσή του αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να γίνει σωστή αξιολόγηση του προηγουμένου του προγράμματος πλαισίου 7 ε, τώρα οι εμπειρογνώμονες παρακολουθούν τι έχει γίνει στο πρόγραμμα πλαίσιο 7 μέχρι τούδε και θα έχουμε την αξιολόγηση στο τέλος του μηνός οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει μία ανακοίνωση αντιδρώντας σε αυτή την αξιολόγηση και από αυτήν θα μπορέσουμε ε, να καταλήξουμε σε ορισμένα συμπεράσματα που θα περιληφθούν για να υπάρξει ε, απλοποίηση όπως έχει προτείνει άρρωστη και η κυρία Καρβάλιο στην εκθεσή της και θα λάβουμε μέτρα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα και για να δείξουμε πώς θα αποδώσει η ε, ημερήσια διάταξη της ε, ε, ε, του στόχου μας. Βλέπω ότι μπαίνουν διάφοροι προσκαλεσμένοι, αλλά θα συνεχίσω με το δεύτερο φλέγον θέμα που είναι ο προπολογισμό, διότι η Επιτροπή παρουσίασε το έγγραφο αναθεωρήσεως του προπολογισμού και αν δείτε θα δείτε ότι η καινοτομία και η ε, έρευνα έχουν μία προεξέχουσα θέση ώστε όχι μόνο τώρα αλλά και στο μέλλον η καινοτομία και η έρευνα να προπορεύονται στην πολιτική ατζέντα όσον αφορά τις ε, δαπάνες και αυτό είναι ένα προήμιο στο πολιετές πρόγραμμα που προβλέπεται για το 2011 ότι θα το καταρτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά πιστεύω ότι και εκεί η θέση μας θα είναι ε, ε, εξέχουσα. Όταν κοιτάμε την στρατηγική του 2020 και τις προσκλήσεις που έχουμε στο θέμα της ενέργειας, ε, της ε, γυράνσεως, ε, της παροχής τροφίμων. Αντιλαμβάνεστε ότι η γενοτομία χρειάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Επίτροπος Φταγιάννη σας είχε παρουσιάσει τις σκέψεις του πρόσφατα. Γι' αυτό και το πρόγραμμα πλαίσιο 8 θα πρέπει να έχει πολύ καλή ισορροπία μεταξύ της έρευνας η οποία θα υποκινείται από την κοινωνία και που αγαπούν οι πολιτικοί σε θέματα όπως η έρευνα στην κύρανση και ούτω καθεξής θα πρέπει ε, συγχρόνως ε, να προωθήσουμε την βιομηχανική έρευνα, να είμαστε ανταγωνιστικοί για την αεροναυτική, για τα φάρμακα, όπου θα πρέπει επίσης να μπορούμε να ηγούμεθα και επίσης θα πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύσουμε στην ε, βάση της επιστήμης, δηλαδή ερευνητική επιστήμη, και εδώ σκέφτομαι με μηχανισμούς όπως το Ερευνητικό Συμβούλιο, οι υποτροφίες και πρέπει να δούμε πώς θα διατυπωθεί αυτό το πρόγραμμα διότι πρέπει να απευθύνεται ή τους πολίτες, να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Γι' αυτό και είμαστε έτοιμοι να καταρτήσουμε ένα πολύ καλό πρόγραμμα μαζί με τους ευρωβουλευτές σε συνεργασία μαζί τους αλλά επίσης οι ενδιαφερόμενοι η επιστημονική κοινότητα. Όλοι θα πρέπει να συμβάλλουν στη διαμόρφωση αυτή. Γι' αυτό και στις 2 Φεβρουαρίου θα παρουσιάσουμε ένα, ένα έγγραφο πολιτικής προσανατολισμού προτού να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε το πρόγραμμα πλαίσιο 8 κατά τρόπον όλοι να έχουμε στοιχεία τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε εις βάθος προτού καταρτήσουμε το πρόγραμμα πλαίσιο 8 το οποίο στη συνέχεια θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο στο τέλος του επομένου έτους. Βέβαια το βασικό μας μέλημα είναι η απλοποίηση. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε αυτό και πρέπει να προχωρήσουμε γι' αυτό και πρέπει να σημειώσουμε και να επιδείξουμε τι χρειάζεται διότι τα μέτρα τα οποία έχετε διαγράψει στην έκθεση σας για τη βιομηχανία είναι πολύ χρήσιμα βέβαια ε, δεν μπορούν όλα αυτά να γίνουν σε λίγους μήνες αλλά ε, την, ε, η πρόθεση σε διάφορα θέματα όπως η, τοκοφόροι λογαριασμοί, η κατάρριξη των τοκοφόρων λογαριασμών, η, στήριξη των μικρομεσών επιχειρήσεων ίσως θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ αλλά να έχουμε υπόψη μας ότι θα υπάρξουν και νέοι κανόνες παιχνιδιού βάση βάσει του προγράμματος 8 διότι το πρόγραμμα αυτό θα διατυπωθεί και θα υποβληθεί μέχρι το τέλος του επομένου έτους όπως είπα για να υποβληθεί στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επίτροπος Γίγαν Queen λοιπόν και εγώ προσπαθούμε να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες για να συνεργαστούμε καλύτερα. Δεν θέλω να σας απασχολήσω υπερβολικά μετά το φαγητό και γι' αυτό θα ολοκληρώσω με λίγα λόγια για το ITER το οποίο έχει συζητηθεί πολλές φορές στην Επιτροπή σας, είναι ακόμη στην ημερήσια διάταξη και θα ήθελα όντως να ζητήσω τη βοήθειά σας για να μπορέσουμε να βρούμε Έχουμε μία λύση για αυτό το πολύ βασικό πρόγραμμα. Πρέπει να επενδύσουμε στο ίτερ και στις μελλοντικές ενέργειες. Δεν έχουμε εναλλακτική λήξη γιατί είναι ένα μέρος του μίγματος και πρέπει να το διερευνήσουμε. Εάν θέλουμε λοιπόν να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα αυτό θα μπορέσουμε να λύσουμε το ενεργειακό που αντιμετωπίζουμε όχι στην Ευρώπη αλλά και όχι μόνο σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπάρχουν πολλά οικονομικά θέματα, διαχειριστικά θέματα και αυτή τη στιγμή ε, βεβαίως πρέπει να διατυπώσουμε σαφείς προτάσεις. Για τα οικονομικά είδατε την πρότασή μας ε, τον Ιούλιο που προτείνουμε 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ προσθήκη για να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτό το πολύ σημαντικό πρόγραμμα και σε επόμενες εβδομάδες θα σας παρουσιάσω ε, μία μια συγκεκριμένη πρόταση για τη διαχείριση του ΙΤΕΡ και τον έλεγχό του για να μπορέσουμε ε, να το υλοποιήσουμε χωρίς να υπερβούμε τον προπολογισμό. Πέραν του 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι πολύ σημαντικό να περιορίσουμε τη συνδρομή πέραν του, του 2,4 στο 1 τρίτον το πολύ, δηλαδή 460 εκατομμύρια και αυτό είναι απαραίτητο διότι το πρόγραμμα πλαίσιο έχει και άλλες προτεραιότητες έρευνα για την υγεία, έρευνα για τη διατροφική ασφάλεια και ως εκ τούτου πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις για το ίτερ αλλά να περιοριστούμε στο 1 τρίτον του συνόλου που χρειάζεται από το 1 1,4 δις και ζητάμε τη βοήθειά σας για το θέμα αυτό. Πολύ σύντομα θα ε, καταλήξουμε σε μία συγκεκριμένη ε, πρόταση για το πόσο θα διαχειριστούμε καλύτερα το ίτερ και θα επανέλθουμε εδώ και από ό,τι ξέρω 9 Νοεμβρίου θα συζητήσετε το ίτερ. Μέχρι τότε θα μπορέσω ενδεχομένως να σας πω πώς θα ελέγξουμε καλύτερα τις δαπάνες ε, γιατί τώρα μετά από εσά θα πάω στο κομπού όπου επίσης συζητούν το ίτερ και θα πρέπει να συζητήσω μαζί τους τις πιο ε, χρηματοοικονομικές πτυχές. Αυτά για να τοποθετήσω το ίτερ στο σωστό πλαίσιο διότι κοστίζει 6,6 δις και υπολογίζεται ότι είναι ε, στην κατανάλωση πετρελαίου μία ημέρας. Δηλαδή το κόστος ε, καταναλώσεως πετρελαίου μίας μέρα είναι το κόστος ολόκληρο του ίτερ για να έχετε σωστή προοπτική του ε, περί τίνος ομιλούμε. Τέλος θα ήθελα να επωφεληθώ, να ευχαριστήσω την κυρία Μάουντ που ήταν μέλος αυτής της Επιτροπής ε, διότι έκανε εξαιρετική εργασία εις ε, την αξιολόγηση ε, και ήταν πάρα πολύ καινοτόμα η πρότασή τους και βρήκαν δυνατότητες να χρηματοδοτήσουν ε, ε, την αξιολογήσουν τη χρηματοδοτική διευκόλυνση καταμερισμού των κινδύνων ε, κατά τρόπον ε, ώστε ε, τα, η, χρηματοδότηση να μην γίνεται άμεσα για την έρευνα αλλά μέσω δανείων και αυτή η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν πολύ καλή και όταν κοιτάω την έκθεση της κυρίας Μαν και του κυρίου Σούτε βλέπω ότι αποφεύγουμε την υπερχρηματοδότηση γι' αυτό και χαίρομαι που η κυρία Μαν ζητά να αποδεσμευτεί η δεύτερη δόση και να αποδοθεί για το πρόγραμμα αυτό και ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα προχωρήσει στην αποδοχή αυτής της προτάσεως για να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση αυτού του μέσου και να έχουμε μία χρήσιμη εφαρμογή των δανείων. Αυτά ήθελα να πω σαν νέος Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας, έρευνας και τεχνολογίας όπως σας είπα διότι από αύριο θα, θα είναι πραγματικό της ήδη η ονομασία. προσβλέπω στη συνεργασία μας και ελπίζω ότι ε, θα συνεργαστούμε πολύ καλά ευχαριστώ σας ευχαριστώ εξ ονόματος όλων των συναδέλφων έχουμε κάποιους συναδέλφους που έχουν ζητήσει τον λόγο και θα σας παρακαλούσα να είστε όσο δυνατόν πιο σύντομοι για να μπορέσουμε να ακούσουμε και κάποιες απαντήσεις. Κυρία Ριέρα Μαδουρέλ πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Σμίθ, να σας καλωσορίσουμε σε αυτή την επιτραπή στην πρώτη σας ε, παρουσία ως ε, νέος Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης ε, Έρευνας και Ανάπτυξης στήξατε πολλά ζητήματα ύψης της σημασίας σε σχέση με το μέλλον της επιστημονικής μας πολιτικής και μερικά από αυτά τα ζητήματα έχουν συζητηθεί σε αυτή την Επιτροπή όπως η απλούστευση και αναμένουμε και την ενδιάμεση αξιολόγηση του 7ου προγράμματος πλαισίου έτσι ώστε να προετοιμάσουμε το 8ο για να δούμε πώς λειτουργήσε επιστημονικά. Καταρχήν το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα από τα ζητήματα που θίξατε και να κάνω και ορισμένα σχόλια ως προς την απλούστευση η κυρία Καρβάλιο, στην οποία αναφερθήκατε, μίλησε για δύο τύπους δράσεων. Καταρχήν την αλλαγή των όρων συμμετοχής και τον δημοσιονομικό κανονισμό, για να δούμε πώς θα εξελιχθούν στο 8ο, 8ο πρόγραμμα πλαίσιο. Υπάρχουν όμως και άλλα μέτρα τα οποία δεν χρήζουν ε, νομοθετικής αλλαγής. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω ποια είναι αυτά τα μέτρα που δεν χρήζουν ε, μετατροπής, δηλαδή νομοθετικών νέων μέτρων πριν αρχίσει το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο. Θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε αυτό το θέμα εκτενέστερα διότι αυτό το θέμα έχει να κάνει με την αύξηση του προϋπολογισμού για το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο. Θα ήθελα να μας πείτε, να μας δώσετε ορισμένα αριθμητικά στοιχεία ή μια ποσοστή αναλογία για να ξέρουμε να έχουμε μια τάξη μεγέθους για την αύξηση πόρων για το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο. Όπως προβλέπετε, θα υπάρξει ανωδική τάση όπως ίσχυσε μεταξύ του έκτου ου και του 7ου προγράμματος πλαισίου. Θα χρειαστούν όμως και άλλες αλλαγές. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε μία ανελικτική πορεία, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν και βαθύτερες αλλαγές πέρα από τα δημοσιονομικά. Μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς προβλέπετε γιατί μιλάμε για αναγκαίες αλλαγές. Τώρα, για, την, ε, για το ίτερ, το ίτερ το έχουμε υποστηρίξει ως πολιτική ομάδα. Αλλά μόλις λάβαμε τη νέα πρόταση για τις ε, δημοσιονομικές προοπτικές και από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν θα αλλάξουν οι προοπτικές και θα αφήσουμε τις μετατροπές για την επόμενη επταετία. Πώς θα χρηματοδοτηθούν προγράμματα τύπου ITER στο μέλλον. Επίσης αναφερθήκατε στον κύριο Βανίστελ Θα πρέπει να δούμε πώς έχει αυτή η συνέργεια μεταξύ προγράμματος πλαισίου και δημοσιονομικών προοπτικών. Πώς ε, μπορούμε να προωθήσουμε μία οριζόντια πειθαρχία. Νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα με την ενδιάμεση αναθεώρηση να, δώσουμε αυτά τα, να μάθουμε αυτά τα νέα στοιχεία. Σε σχέση τώρα με αυτό, αυτή τη χρηματοδοτική διευκόλυνση καταμερισμού των κινδύνων, το RSFF λειτουργήσε ικανοποιητικά θα δούμε τι θα μας πούν η, κυρία Μάν και ο κύριος Σέτε, αλλά επειδή είσαστε παρόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο αυτό το μέσον λειτουργήσε καλά. Δηλαδή τα προγράμματα ευρείας κλίμακας ε, βρήκαν ανταπόκριση σε αυτό το RSFF υπάρχουν και προγράμματα μεγαλύτερου κινδύνου που θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Σε ποια προγράμματα λειτουργήσε καλύτερα δηλαδή αυτό το χρηματοοικονομικό μέσο καταμερισμού των κινδύνων. Υποθέτω ότι αυτά θα μας τα προσδιορίσουν καλύτερα οι συντάκτες της έκθεσης, αλλά νομίζω ότι και εσείς μπορείτε να βοηθήσετε σε αυτή τη διαδικασία. Η κυρία Καρβάλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Γενική Διευθυντά. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Πρώτα απ' όλα, να σας ευχαριστήσω για την καλή συνεργασία που είχαμε και με εσάς και με την υπηρεσία σας για την έκθεση απλοποίησης. Η έκθεση είναι απλά η αρχή. Τα δύσκολα είναι αυτά τα οποία έρχονται, δηλαδή η εφαρμογή και βεβαίω αυτό είναι μια διαδικασία περιπλοκή και δύσκολη και προβλέπω πως θα βρείτε κάποια εμπόδια ε, για να μπορέσετε να εφαρμόσετε αυτά τα οποία περιέχονται στην έκθεση και στην ανακοίνωση. Έχουμε βεβαίω εμπιστοσύνη στο ρεαλισμό σας και στις ηγετικέ σας ικανότητες και στον Επίτροπο που υποστηρίζει το θέμα αυτό και βεβαίω εμείς θέλουμε η απλοποίηση να είναι στο προσκήνιο όπως μας ζητήσατε για να μπορέσετε να ξεπεράσετε τα εμπόδια τα οποία θα συναντήσετε για την εφαρμογή του προγράμματος αυτού. Θα ήθελα να σας ζητήσω να είστε πιο συγκεκριμένος όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Υπάρχουν μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα, είναι κοινή λογική, δεν χρειάζονται καμία αλλαγή στους κανονισμούς. Υπάρχουν κάποια άλλα τα οποία θα εισαχθούν με την ανθεώρηση του 7ου προγράμματος πλαισίου και άλλα στο 8ο πρόγραμμα πλαίσιο. Όσον αφορά δε, το κόστος προσωπικού υπάρχει πολλή πίεση από πλευράς ε, ερευνητών για να ξεκινήσετε να το εφαρμόζετε αυτό και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν, μπορεί, αν βλέπετε κάποια εμπόδια εκεί πέρα και το τι μπορούμε να κάνουμε. Το δεύτερο ερώτημα αφορά το ITER πώς μπορούμε να έχουμε εγγυήσεις πως η τωρινή κατάσταση δεν θα επαναληφθεί. Γιατί ελπίζουμε να λυθεί η τωρινή κατάσταση, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε πως κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί, γιατί, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η κατάσταση δεν οφείλεται σε απρόβλεπτα επιστημονικά αποτελέσματα, είναι περισσότερο θέμα δομών και διαχείρισης ή έλλειψης διαχείρισης. Όσον αφορά δε το μέσο διαμερισμό του κινδύνου, αντιλαμβάνομαι πως κάποια μικρομεσαία κράτη δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό και έχουν πρόσβαση σε αυτά τα έργα. Αν μπορέσετε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες και από αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Τσουκαλάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ευτυχής να υποδάχομαι τον κύριο Σμίτς στην Επιτροπή. Με άλλη ιδιότητα είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί, μου, μαζί του και έχω τις καλύτερες εντυπώσεις και έχω μεγάλες ελπίδες όπως όλοι μας για το έργο που πρόκειται να επιτελέσει εδώ. Ο κύριος Σμίτς ε, έχει μια πολύ καλή αντίληψη γιατί συμμετείχε σε όλες τις κύριες δράσεις από την ΕΡΑ μέχρι το ΚΟΣΤ και από το ΕΣΦΡΙ μέχρι την ΕΖΑ και επομένως ξέρει πολύ καλά το χώρο. Υπό αυτή την έννοια εγώ θα ήθελα να εστιαστώ πρώτον σε μία μόνιμη απορία που όπως ξέρετε κύριε Πρόεδρε τη διαπιστώνω πάντοτε θα ήθελα να μας πει ο κύριος Σμιτς εάν έχει μια συγκεκριμένη ε, γνώση για το τι ακριβώς κάναμε με τη στρατηγική της Λισαβόνας. Θα ήθελα να ξέρω δηλαδή σε τι αντιστοιχεί η προφητεία μας, το όραμά μας του 2000, ότι το 2010 θα είμαστε η πιο ανταγωνιστική οικονομία παγκόσμια, βασισμένη στην οικονομία της γνώσης, και ποιες είναι αυτές οι προοπτικές. Εάν δεν ξέρω, δεν έχω απαντηθεί ή δεν μου έχει πει κανείς τι συνέβη με αυτή τη στρατηγική, και κατά πόσο βλέπω τώρα ότι έχουμε ένα νέο όραμα, το όραμα 2020, ε, ξέρω από την ψυχιατρική ότι υπάρχουν τριών ειδών οράματα. Το όραμα που έχει ένας που στηρίζεται στην πραγματικότητα και προβλέπει το μέλλον, το όραμα ενός προφήτη, το όραμα ενός ποιητή και το όραμα ενός φρενοβλαβούς. Θα ήθελα επομένως να έχω συγκεκριμένα πράγματα για αυτά τα οράματα που συνεχώς βάζουμε. Για παράδειγμα, από ε, παρακολούθηση παρουσιάσεων που έχετε κάνει στο παρελθόν καταλαβαίνω ότι ε, διάφορες δυσκολίες που είναι δομικού τύπου ε, τις επισημαίνετε και εσείς ο ίδιος. Για παράδειγμα, σε μια παρουσίασή σας που κάνατε για το αέρα, παρατηρείτε ότι το 75% της παγκόσμιας επένδυσης σε έρευνα είναι έξω από την Ευρώπη. Παρατηρείτε ότι μειώνεται η συμμετοχή μας στο νέο τοπίο το παγκόσμιο σε S&P. Ε, Παρατηρείτε ότι έχουμε μια stagnation στην ένταση του R&D στην Ευρώπη ενώ αυξάνεται της Ασίας. Παρατηρείτε ότι έχουμε χαμηλή ένταση ιδιωτικών επενδύσεων σε R&D στον ιδιωτικό τομέα. Υπό την έννοια αυτή, ενώ όλα τα πράγματα τα οποία λέμε εδώ είναι πολύ σπουδαία, ναι θέλουμε αυλοποίηση θέλουμε, θέλουμε, θέλουμε, εγώ θα ήθελα να δω με μεγαλύτερη ευκρίνεια τι ακριβώς μπορούμε να περιμένουμε το 2020, διότι το Global Trends in 2025 μου δείχνει ότι τα πράγματα θα γίνουν ε, ακόμα πιο δύσκολα για την Ευρώπη ε, αν βάλει κανείς μέσα και την κρίση, αν βάλει κανείς την άνοδο των BRIC, αν βάλει το μεγάλο χάσμα μεταξύ της καινοτομίας ε, ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία για παράδειγμα, μια που τώρα είστε και θεσμικά υπεύθυνος και για την καινοτομία και μια που σύμφωνα με έναν ορισμό η έρευνα είναι η μετατροπή χρήματος σε γνώση και η καινοτομία είναι η αντίστροφη, δηλαδή η μετατροπή της γνώσης σε χρήμα, τότε έχουμε πρόβλημα αν δεν συμβαίνει αυτός ο κύκλος στο τρίγωνο της γνώσης. Ανησυχώ πολύ για το γεγονός ότι μολονότι έχουμε κατά μέσο όρο καλύτερα πανεπιστήμια από τα Αμερικάνικα, δεν έχουμε τα καλύτερα, δεν πλασαριζόμαστε καλά στα extremes, στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου και συνεπώς μου είναι αδιάφορο εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση παράγει περισσότερες επιστημονικές δημοσιεύσεις αφού στις καλύτερες δημοσιεύσεις το ποσοστό της είναι πολύ φτωχότερο από τον άλλον. Με αυτή την έννοια θα ήθελα δομικά να μου πείτε ποιο είναι το δικό σας όραμα για την Ευρώπη του 2020 και πόσο ρεαλιστικά είναι αυτά τα μεγάλα λόγια που λέμε. Επειδή προέρχομαι μια, από μια χώρα που τα μεγάλα λόγια συνήθως πληρώνονται με μεγάλες τιμωρίες, θα ήθελα να δω μπας και μας συμβεί και τίποτα τέτοιο εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Χατζημαρκάκης. Ναι, άκουσα με ευχαρίσει αυτά τα οποία είπε ο κ. Τσουκαλάς. Πρώτα απ' όλα σας συγχαίρω και εύχομαι καλή επιτυχία στη σας ως ε, γενικός διευθυντής σε ένα πάρα πολύ σημαντικό τομέα. Λοιπόν, ας δούμε λίγο. JRC, ERCIT, ε, πρόγραμμα 7, JTI, MISIP κτλ. Τεχνολογική πλατφόρμα και τώρα βρήκατε άλλο ένα αρκτικό λέξο το Innovation Partnerships. Να σας πω, ως βουλευτής που ασχολούμαι με αυτά τα θέματα, που έχω αρμοδιότητα γι' αυτά, ε, κάποια στιγμή έχει αρχίσει και με ενοχλεί. Δηλαδή, έχουμε διάφορα πλαίσια, γραμμές, πολλές φορές ε, επικαλύψεις και μπορώ να σας πω άρα πως και η προσέγγιση μας, την οποία ανέφερε η κυρία Καρβαλιό και την οποία επεξεργαστήκαμε όλη στην έκθεση αυτή, Δηλαδή η προσέγγιση μόνο με την απαρίθμηση όλων αυτών που σας είπα γίνεται κάτι το παράλογο. Συγκεκριμένο ερώτημα τώρα. Ορίστε μου ένα έργο ορόσημο το οποίο μπορώ να πω σε κάποιους ότι στους ψηφοφόρους μου να ότι κάνουμε αυτό το έργο το ευρωπαϊκό. Ούτε το ίτερ είναι αυτό, ούτε ο γιατί έχουν μάλλον αρνητική εικόνα αυτή τη στιγμή. Και μιλάμε για ακόμη περαιτέρω, ακόμη περαιτέρω κατακαιρματισμό του τοπίου της έρευνα, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αντέξουμε, δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Εν τω μεταξύ μιλάμε για 50 δισεκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον στο πρόγραμμα 7. Θα ήθελα καλό τουλάχιστον να ξέρουμε πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά για να αποφεύγουν οι αλληλεπικαλύψει κάτι το οποίο δεν γίνεται γιατί δεν υπάρχει βάση δεδομένων. Οπότε θα πρέπει τουλάχιστον αυτό να εγγυηθούμε, δηλαδή να μην υπάρχει αλληλεπικάλυψη, να κάνουμε δύο φορέ την ίδια δουλειά και δεύτερον κάποια μεγάλα έργα, ορόσημα, τύπου να στείλουμε κάποιο στο φεγγάρι, αλλά να μπορέσουμε να τα πούμε στου ψηφοφόρου μα ότι κάνουμε αυτή την, ε, αυτό το το έργο. Ο Νίξον πριν από 30 χρόνια είπε θέλω να καταπολεμήσω τον καρκίνο, να τον νικήσω. Δεν τα κατάφερα, αλλά πάρα πολλά από τα έργα που ξεκίνησαν στην έρευνα αυτή κατά του καρκίνου βοηθούν πάρα πολλούς ανθρώπους. Εμείς δεν έχουμε τέτοια στόχευση, τη χρειαζόμαστε. Έχετε μια ιδέα τι, ποιος θα μπορούσε να είναι ένα τέτοιο στόχος τώρα για το ίτερ. Να σας πω ξεκάθαρα, σας άκουσα, άκουσα αυτό το οποίο είπατε, I hear you στα αμερικανικά, αλλά θα ήθελα να πω πως είναι κρίμα και βαρέστηκε αυτό το κοινοβούλιο να ακούει πως τα κράτη-μέλη και οι Κομισιόν δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν σωστά τα έργα. Εμείς ως α, ελεγκτές του υπερβολογισμού που είμαι και εγώ θέλουμε να ξέρουμε τι γίνεται εδώ πέρα. Να σου πω, είναι απλό. Εμείς ως Ευρωπαίοι πληρώνουμε το πενταπλάσιο από τους Αμερικάνους, Ιαπωνέζους για το ίτερ λάβαμε την έδρα για αυτό το λόγο. Εάν είχαμε και πέντε φορές το λέγειν των υπολείπων, δεν θα υπήρχε ένα πρόβλημα. Αλλά δεν συμβαίνει αυτό, ανταυτού μόνο πληρώνουμε. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να αλλάζει η ουσία άλλων προγραμμάτων όπως το CP το 7ο πλαίσιο μόνο και μόνο για να μπορούμε να συνεχίζουμε άλλα 30 χρόνια να πληρώνουμε το ίτερ και θα επιτύχουμε κάποιο αποτέλεσμα σε 30 χρόνια. Δεν γίνεται έτσι. Και σας έχω πραγματικά καλή τύχη με όλα αυτά. Λοιπόν, έχω ακόμη πέντε συναδέλφους ε, τους οποίους ακούσουμε και μετά τις απαντήσεις και Τέσσερις ώρα τέλος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, πολύ σωστά έρχομαι μετά τον κύριο Χατζημαρκάκη διότι και εγώ στηρίζω αυτή τη συγχώνευση αλλά θα πρέπει να υπάρξει λογική διαχείριση και λογικές προτάσεις διότι διαφορετικά δεν θα τα βγάλουμε πέρα. Ευχαρίσω να αγωνιστούμε και για άλλα προγράμματα δεν θέλω να επισέλθω στο Γαλιλαίο διότι υπάρχουν διάφορες συζητήσεις δεν είναι ε, θέμα της, ε, της αλλά των κρατών μελών και των ε, επιχειρήσεων που συμμετέχουν. Θα ήθελα όμως οι μικρομεσαίες επιχειρήσει να μπορούν να χαρούν διότι ερευνούμε και για λογαριασμό τους και μιλάμε για απλοποίηση. Περιμένουμε ένα γωνίο στο πρόγραμμα πλαίσιο 8, αλλά έχω ακούσει ότι είναι δύσκολο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντεπεξέλθουν με τα μικρά κονσόρτσια. Οπότε ε, τι λέτε εσείς, έχετε ακούσει κάτι επ' αυτού ή μπορούμε να ρωτήσουμε κάποιον συγκεκριμένα αν σωστά υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες. Ευχαριστώ. Κύριε Γενικέ Διευθυντά, κύριε Πρόεδρε, όλοι ε, έχουν εκφραστεί επί του θέματος επαρκώς. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι μιλάμε για έρευνα και ανάπτυξη για αυτό το ευρύτατο κεφάλαιο για το οποίο φέρουμε μεγάλη ευθύνη. Εκτός αυτού όλοι μιλάνε, οι πολιτικοί, οι βιομήχανοι, ο μέσος πολίτης, όλοι έχουν κάτι να πούν και το βλέπουμε παντού. Εγώ νομίζω ότι θα επιλύσουμε το θέμα της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας αν κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση όχι με λόγια αλλά με πράξεις. Γιατί τώρα θα πρέπει να τεθεί το θέμα πραγματικά επιτάπητος. Είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Σήμερα στην Ολομέλεια γίνεται λόγος για τον ουρανό και τον κυβερνοχώρο, για τους δορυφόρους, για την ανάπτυξη, για την έρευνα και πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε μία μεγάλη όθηση στο θέμα αυτό. θα πρέπει να δούμε αν θα πρέπει να γίνουν άρδιν αλλαγές. Και επιμένω, επειδή αρχίσαμε αυτή την πολιτική με το ίτερ, διότι η ενέργεια με βάση τη σύνδεξη είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα συνοδευτικό πρόγραμμα για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε αυτές τις δοκιμές ίτερ και να υπάρχει μία σωστή διακυβέρνηση, διότι είναι ένα πολύ περίπλοκο πρόγραμμα. Εύχομαι να τα καταφέρουμε. Ελπίζω να μπορέσετε να αρχίσετε με αυτή την εργασία που είναι ύψης της σημασίας για το μέλλον μας. Ευχαριστώ. Κύριε Σμίτς, και εγώ θέλω να σας συγχαρώ για τον καθορισμό σας. Ε, νομίζω ότι ε, τα νέα φαίνονται ε, καλός ιονός αλλά πρέπει να ασχοληθούμε με τα ουσιαστικά θέματα. Όσον αφορά την έρευνα και την ε, καινοτομία, ακούμε για την καινοτομία αλλά μέχρι στιγμής τα σχόλια της Επιτρόπου υπήρξαν ασαφή. Έχουμε νέο όνομα αλλά τον παλιό προϋπολογισμό, το πρόγραμμα πλαίσιο και γι' αυτό πρέπει να αντιληφθούμε τι σημαίνει η καινοτομία και τι μετακινήσεις προβλέπονται δημοσιονομικά. Όσον αφορά το SRF ποτέ δεν το απορρίψαμε αλλά σχετικά με την χρηματική διευκόλυνση καταμερισμού των κινδύνων θα ήθελα να ξέρω ποιο βάρος θα έχει. Το αξιολογούμε θετικά αλλά ε, υπάρχει ένα παράδειγμα δηλαδή ε, ε, θα υπάρξει έρευνα και θα χρηματοδοτήσετε βιομηχανικά προγράμματα είναι ένα μέσο ή είναι ένα παράδειγμα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε για να δούμε που θα καταλήξουμε. Όσον αφορά το ίτερ, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, το ΕΛΚ έχει καταρτήσει ένα έγγραφο σχετικά με το ίτερ, σχετικά με τη δομή διαχείρισης κτλ. Από τις 7 Νοεμβρίου και μετά δεν θα ασχοληθούμε εμείς, αλλά οι δημοσιονομικοί μας συνάδελφοι που θα συζητήσουν τη χρηματοδότηση του ίτερ και καλό θα ήταν να έχουμε συμφωνήσει στα διαρθρωτικά θέματα και ο πρόεδρος πριν ξεκινήσει η διαδικασία προϋπολογισμού να λάβει επί του θέματος ένα γράμμα διότι διαφορετικά θα βρούμε μια δημοσιονομική λύση η οποία δεν θα είναι αναγκαστικά και πολιτική. Το θέμα που έθεσε ο συνάδελφος Χατζημαρακάκης με ενδιαφέρει ιδιαίτερος, ο GRC, διότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλει τώρα να έχει έναν σύμβουλο σαν αυτόν που ε, έχει από καιρού ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έναν επιστημονικό σύμβουλο και το ερώτημα είναι τι σημαίνει αυτό για, τον, για τη γενική σας διεύθυνση Δηλαδή αυτό θα είναι αποσπασμένος εις, ε, την, ε, εις τον πρόεδρο ή τις σχετικές συζητήσεις θα τις κάνει η Επίτροπος. Θα είναι ένα συμβουλευτικό όργανο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι διάφορα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν ταχύτατα. Μετά, τα SME. Πρέπει να είμαστε ειλικρινεί όταν συζητάμε το θέμα αυτό, διότι από τη μια μεριά ζητάμε μεγάλα προγράμματα και από την άλλη πλευρά βέβαια όταν αυτά τα μεγάλα ε, τα μέσω, μέσου μεγέθους προγράμματα είναι κατάλληλα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να δούμε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε και πού να πετάξουμε τα δικά μας τα φτερά διότι ε, θα πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη κατάρτιση των προγραμμάτων γιατί αν θέλουμε μεγάλα προγράμματα δεν μπορούμε να επιβαρύνουμε με αυτά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να τους ζητήσουμε να, τις, ε, να τα προωθήσει. Ο κύριος Περίλο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω εντάχει να παρέμβω, διότι ο Γενικός Διευθυντής έχει ε, διοριστεί τώρα πρόσφατα και από αύριο αρχίζει το πραγματικό του έργο. Θα ήθελα να του πενθυμίσω ότι μας απασχολούν δύο ε, ευρύτατα ζητήματα. Το ένα είναι το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και το άλλο το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο. Θα πρέπει να βασιστούμε στις δυσκολίες του 7ου προγράμματος πλαισίου και αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης και σε αυτή την Επιτροπή. Δύο επισημάνσεις θα ήθελα να κάνω. Επειδή θα πρέπει να απομακρυνθούμε από το παρελθόν, επειδή ακριβώς δεν απέδωσε, δεν έφτασε στα επιθυμητά αποτελέσματα, αυτή ακριβώς θα πρέπει να είναι η κατευθυντήριά μας γραμμή θα πρέπει να ασχοληθούμε με την απασχόληση. Αυτό είναι το σημείο εκκίνησης και για την έρευνα και καινοτομία. Αλλά ο βασικός στόχος είναι τα αποτελέσματα της έρευνας που θα πρέπει να δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης. Εδώ θα πρέπει να... Αυτό το ζήτημα πρέπει να μας απασχολήσει πολύ περισσότερο. Τέλος ως προς την απλούστευση θα ήθελα να πω ότι η απλούστευση βοήθησε στην ανάπτυξη της Ευρώπης. Είναι ιδιαίτερα δεσμευτική εργασία και βεβαίως υφίσταται μεγάλη δοκιμασία το ολοπλαίσιο εργασίας, γι' αυτό σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Λάμπερτς. Ναι κύριε Πρόεδρε. Λόγω διένειας δεν θα κάνω κάποια ερώτηση γιατί πρέπει να φύγω να πάω να ψηφίσω σε πέντε λεπτά. Οπότε νομίζω κύριε Διευθυντά καλύτερο είναι να συζητήσουμε τις ερωτήσεις που έχω τέτα τέτ, γιατί δεν θα μπορέσω να ακούσω την απάντηση. Σπάνιο αυτό το οποίο κάνετε. Σας ευχαριστώ, ναι. Ναι, ναι, όχι, είναι σωστό. Κύριε Γενική Διευθυντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας και τα σχόλιά σας. Νομίζω πως η κυρία Μαδουρέλ σωστά έθεσε επιτάπητος ε, την απλούστευση, κάτι το οποίο είναι πολύ ψηλή προτεραιότητα δική σας και δική μου και σχετίζεται και με το ερώτημα της κυρίας Καρβάγιο, τι μπορούμε να περιμένουμε τώρα και τι αργότερα. Στόχος μας ως ε, έτσι, γρήγορο όφελος και χωρίς να χρειαστεί να αλλάξουμε το νομικό πλαίσιο είναι πως εξετάζουμε αυτή τη στιγμή, βεβαίως αυτά είναι ακόμα σκέψεις, να εισαχθεί αυτό το μέσο κόστος προσωπικού, να δούμε τι θα γίνει με το ζήτημα των λογαριασμών των τοκοφόρων, κατά αποκοπήν ποσά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βεβαίως να εισαχθούν διατάξεις για εναρμονισμένη ερμηνεία κανόνων και διαδικασιών. Γι' αυτό το τελευταίο σημείο στο οργανόγραμμα το νέο της Γενικής Διεύθυνσης το οποίο θα κριθεί αύριο από το Σώμα των Επιτρόπων ακριβώς στόχο έχουμε ένα οργανόγραμμα το οποίο σημαίνει πως θα υπάρχει ενιαία ερμηνεία των κανονισμών ε, και των διαδικασιών σε όλες τις υπηρεσίες κομισιών. Και τα άλλα μέτρα θα υποβληθούν ελπίζω μέχρι τα Χριστούγεννα και οτιδήποτε απαιτεί βεβαίω τροποποίηση των κανόνων συμμετοχής που είναι η διαδικασία συναπόφασης όπως ξέρετε όπως παραδείγματος χάρη η εισαγωγή των αρχών λογιστικής ε, των συμμετεχόντων θα πρέπει να περιμένει μέχρι το 2011 όταν θα υποβάλουμε προτάσεις για τους νέους κανόνες συμμετοχής. Η κυρία Μαδουρέλ επίσης ανέφερε τον προπολογισμό του πλαισίου προγράμματος 8, είπατε πως θέλετε υψηλότερο προπολογισμό. Η δήλωσή μου ήταν πως σημείωσα και στα έγγραφα 2020 και στην αναθεώρηση του προπολογισμού πως η έρευνα και η καινοτομία είναι πρώτη προτεραιότητα. Μιλάμε δηλαδή για να γίνουν τα πράγματα ξυπνότερα και πιο πράσινα. Οπότε μιλάμε για καινοτομία. Το εάν θα λάβουμε βέβαια περισσότερα κονδύλια είναι άλλη υπόθεση. Ελπίζω ναι, αλλά βεβαίως όλα αυτά περνάνε από τα δικά σα χέρια ω αρχή του προπολογισμού μαζί με το Συμβούλιο, με τα κράτη-μέλη. Αλλά εάν θέλουμε να έχουμε μια οικονομία τη γνώση στην Ευρώπη, πρέπει να επενδύσουμε σε αυτήν. Βεβαίως, το ΙΤΕΡ, ένα ζήτημα που το αναφέρατε όλοι, εγώ διορίστηκα 1η Ιουλίου, από την πρώτη μέρα αντιμετώπισα το ίτερ. Πρώτα απ' όλα σκοπεύω να λύσω το ζήτημα του προϋπολογισμού. Έκανα πρόταση για τα επιπλέον 1,4 δισεκατομμύρια. Ελπίζω να ξεκαθαρίσω το ζήτημα γρήγορα συνδιαλλαγή. Τώρα, αν θα έχουμε περαιτέρω υπερβάσεις του κόστους. Όχι όσο είμαι εγώ γενικός διευθυντής. Αυτό δεν θα το δεχτώ και ο Επίτροπος είπε ξεκάθαρα πως δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Όσον αφορά τώρα την διαχείριση, πώς θα μπορέσουμε να περιορίσουμε το κόστος και να διασφαλίσουμε αναθεώρηση της ε, διακυβέρνησης. Θα καταθέσουμε σύντομα, θα υποβάλουμε σας σύντομα προτάσεις και στο Συμβούλιο Υπουργών, αλλά ήδη έχουν γίνει κάποιες αλλαγές σημαντικές αλλαγές. Γνωρίζετε πως και ο Γενικός Διευθυντής ε, του ΙΤΕΡ απομακρύνθηκε από τη θέση του, όπως επίσης ε, και ο Διευθυντής ε, στην Βαρκελόνη απομακρύνθηκε από την θέση του. Οπότε έγιναν δραματικές κινήσεις για να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν θα είναι απλά πολιτικοί διορισμοί, αλλά θα μπορούν να διαχειριστούν την κατάσταση. Όμω, πρέπει οι άνθρωποι να ξέρουν τη δουλειά του και να μπορούν να κάνουν τη δουλειά του. Επίση, αναφερθήκατε στο RSFF, δεν θα πω περισσότερα πράγματα εδώ πέρα, γιατί και έργα είναι εδώ πέρα. Πράγματι, το RSFF είναι μεγάλο για έργα βιομηχανικά μεγάλη κλίμακα. Βεβαίω είναι πολύ πολύπλοκο για μικρομεσαίες επιχειρήσει και αυτό σχετίζεται και με τις ιδιαιτερότητες ε, αυτού του target group που είναι μικρό και δύσκολο στο να το πλησιάσουμε, αλλά προσπαθήσαμε να βρούμε κάποιου καινοτόμου τρόπου για να προσεγγίσουμε ομάδε μικρομεσαίων επιχειρήσεων, π.χ. δόθηκε στο Eindhoven στην Ολλανδία σε ένα επιχειρηματικό πάρκο που βρίσκεται εκεί πέρα σε μια ομάδα επιχειρήσεων ένα δάνειο και είμαι εντυπωσιασμένο από τα πρώτα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται έτσι. Η ιδέα, κυρία Καρβάγιο αναφέρθηκε στην απλοποίηση, αναφέρθηκα ήδη στο ερώτημά σας τι θα κάνουμε γρήγορα και τι θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Επίσης, για το RSFF, είδαμε πως ε, παρά το ότι είναι ένα νέο μέσο, ε, ότι υιοθετήθηκε γρήγορα, ήδη εκταμιέθηκαν πάρα πολλά δάνεια, αλλά και σε πάρα πολλά κράτη-μέλη και σε συνδεδεμένες χώρες, από το Ισραήλ, την Τουρκία, από κράτη-μέλη στην ε, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία. Οπότε σταδιακά ανεβαίνει ο ρυθμός, αλλά υπάρχουν βεβαίως κάποιες ε, στενοποί και σωστά είπατε πως θα πρέπει να ξεκαθαριστεί και το ζήτημα και να ληφθούν κάποια διορθωτικά μέτρα. Ανέφερα επίσης πως θα δούμε το ζήτημα Twitter για να μην έχουμε πάλι υπερβάσεις του κόστους όσο είμαι εγώ γενικός διευθυντής την ίδια άποψη και ο Επίτροπος. Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε στρατηγική της Λισαβόνας και είπε πώς διαφέρει από τη νέα στρατηγική και γιατί απέτυχε. Κατά την άποψή μου, η στρατηγική της Λισαβόνας ήταν επιτυχία σε μεγάλο βαθμό, γιατί ήταν μια στρατηγική η οποία ε, είχε ψηλά στι προτεραιότητε στην έρευνα και την καινοτομία. Και βέβαια, εντάξει, η Ευρώπη δεν έγινε το 2010 η πιο ανταγωνιστική οικονομία του κόσμου, δεν το επιτύχαμε αυτό, αλλά ε, επιτύχαμε μεγάλη πρόοδο όσον αφορά το να αποκτήσει σημασία η έρευνα και η καινοτομία. Μία από τις αποτυχίες, αποτυχίες ε, της στρατηγικής Λισαβόνας ήταν ότι δεν το είδαν ως κάτι δικό του τα κράτη-μέλη. Το είδαν ως κάτι των Βρυξελών. Γι' αυτό νομίζω πως η στρατηγική Ευρώπη 2020, την οποία τη συζητήσαμε ευρύτατα μαζί σας, με τα κράτη-μέλη ε, είναι κάτι το οποίο το βλέπουν ως κάτι δικό τους τα κράτη-μέλη και έχει πιθανότητες επιτυχίες. Αλλά για να είμαι σαφής, αν μιλάμε για τις δαπάνες στον τομέα αυτών, τα κράτη-μέλη πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνε τους. Έχουν το 95% της χρηματοδότησης και Βεβαίω η Ευρώπη θα είναι ισχυρή στην έρευνα και την καινοτομία μόνο εάν εμπλακούν και τα κράτη-μέλη. Και βλέπουμε κάποια καλά παραδείγματα κρατών μελών παρά την κρίση επενδύουν στην οικονομία τη γνώση, Αν δούμε τη Γερμανία, το 2011 θα ξοδέψει 11 δισεκατομμύρια σε έρευνα και καινοτομία. 7,2 παραπάνω σχέση με το 2010 και 54% σχέση με το 2005 και σκοπεύει να φτάσει το στόχο του 3% τα επόμενα δύο χρόνια. Οπότε, όπως σας είπα, η οικονομία της γνώμης θα έχουμε μόνο εάν επενδύσουμε σε αυτήν. Και υπάρχουν και κάποιες σκανδιναβικές χώρες που είναι διατεθειμένες να το κάνουν. Και δεν επενδύουμε μόνο εμείς. Η Σιγκαπούρη είναι στο 5%. Η Κίνα τα αυξάνει, αυξάνει τις απάνες κατά 22% το έτος, οπότε αυτό δεν είναι κάτι που είναι μόνο δική μας προτεραιότητα, αλλά και στην Άπο Ανατολή. Βεβαίω στην Άπο Ανατολή δεν το λένε. Μόνο τα κάνουν κιόλα, επενδύουν κιόλα, ενώ στην Ευρώπη δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πράγματι έχει δίκιο ο κύριο Τσουκαλά, πρέπει να κάνει και ο ιδιωτικός τομέα περισσότερα. Εδώ πέρα η Ευρώπη είναι πίσω σε σύγκριση με τη ΣΥΠΑ και την Ιαπωνία και οι ιδιωτικές επενδύσεις πρέπει να αυξηθούν. Ο κύριο Χατζαμαρκάκη έχει δίκιο, υπάρχουν πάρα πολλά μέσα. Ένα δάσος ολόκληρο και πρέπει, ότι πρέπει να το αναθεωρήσουμε τελείως. Το ανέφερε και η κυρία Καρβάλιο στην έκθεσή της. Πρέπει να φύγουμε από αυτή τη σύγχυση που επικρατεί στην επιστημονική κοινότητα και στις βιομηχανίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Σκοπεύουμε οπωσδήποτε να το κάνουμε και κάποια από αυτά τα με κοπούν αναφέρατε τα έργα μας τα οποία θα μπορούσαν να είναι ορόσημα. Εγώ θα ήθελα να έχω αυτό το ζήτημα της, γύρα, της υγιεινής γύρανσης. Το Alzheimer είναι τεράστιο ζήτημα για την κοινωνία μας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 1% και είναι η πρώτη φορά στην ιστορία, 1% είναι το κόστος, 1% του ΑΕΠ, είναι το κόστος ε, του Alzheimer. Και βεβαίως πέρα από το ανθρώπινο κόστος υπάρχει και το οικονομικό εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα έργο που πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, κράτη-μέρη, κομισιόν, περιφέρειες, να ε, αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Εάν δείτε την έρευνα περί Αλτσχάιμερ αυτή τη στιγμή, είναι κατακαιρματισμένη. Υπάρχουν εκατοντάδες εθνικά και περιφερειακά προγράμματα χωρίς καμία κλίμακα και σπαταλάμε χρήματα. Και αυτό το οποίο με συναρπάζει, όταν ενώνεται η Ευρώπη, αν δείτε το Airbus, το CERN, είμαστε οι καλύτεροι στον κόσμο και μπορούμε να ανταγωνιστούμε τους πάντες. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό και στην έρευνα για το Alzheimer. Θα επενδύσουμε σε αυτό πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια. Πρόγραμμα πλαίσιο 8. Πράγματι πρέπει να γίνει σοβαρός έλεγχος και αξιολόγηση δικτύπου εξ άντε. Για κάθε ευρώ θα δώσουμε λογαριασμό και σε εσάς και στο Συμβούλιο και στον φορολογούμενο και θα κάνουμε μόνο πράγματα που έχουν ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Το και πάλι έχετε δίκιο κύριε Χατζημαρκάκη, υπάρχουν προβλήματα. Προσπάθησα να αναλάβω μέτρα για να αρχίσουμε να προχωράμε. Δεν μπορούμε παρά να επενδύσουμε στο ίτερ, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Πρέπει να σφίξουμε τα δόντια όσον αφορά την ε, χρηματοδότηση, όσον αφορά το θέμα της διακυβέρνησης και της διαχείρισης και θα καταθέσουμε προτάσεις. Έχετε δίκιο στο θέμα της διακυβέρνησης είναι περιορισμένη η ψήφος της κοινότητας ενώ δίνουμε τα περισσότερα λεφτά. Κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε. Το σχόλιο του κυρίου Γκλάντε κατόπιν για τη σύνδεξη και πάλι έκανα την σχετική δήλωση. Πράγματι χρειάζεται καλή διαχείριση εδώ πέρα. Μικρόμεσες επιχειρήσεις, ναι, σωστά, είναι σημαντικό μέρος του στόχου του προγράμματος πλαισίου. 50% των δαπανών έχουμε αφιερώσει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κύριο Σέιλε, σωστά ανέφερε πως πρέπει να κάνουμε μία επιλογή. Εάν θέλουμε να επιλέξουμε μεγάλα προγράμματα ή εάν θέλουμε να ασχοληθούμε με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Πρέπει να κάνουμε επιλογές, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Κάντσιαν, Πράγματι η σύνδεξη είναι κάτι το ελκυστικό. Χαίρομαι που μας στηρίζετε. Χρειαζόμαστε εδώ πέρα καλύτερη διακυβέρνηση. Και τέλος, για να τελειώσω με τον κύριο Έιλερ, λέει σαφώς ο επιστημονικός σύμβουλος. Ναι, ο Μπαρόσο είπε πως θα ορίσει έναν επιστημονικό σύμβουλο. Και είναι φανταστική ιδέα. Είναι πολύ καλή ιδέα διότι ο κύριος Μπαρόζο αυτή τη στιγμή έχει το έγγραφό του, έχει οικονομολόγους γύρω τους και ε, θέλει μεταξύ των προσωπικών συμβούλων του να έχει και έναν επιστήμονα. Θέλει να μπορεί να παίρνει ε, πολιτικές αποφάσεις οι οποίες έχουν ε, επιπτώσεις επιστημονικές και αυτός ο επιστήμονας θα πρέπει να συνεργάζεται ένα με το κέντρο έρευνας. Και τέλος, κυρία Πυρίλο, όσον αφορά το πρόγραμμα πλαίσιο 7, πρέπει να καταλήξουμε σε συμπεράσματα κατά τρόπον ώστε να διαμορφώσουμε το πρόγραμμα πλαίσιο 8 σε συνεργασία μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Σμιτ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι πολλές ευχές και όσον αφορά την πρόταση για το ΙΤΕΡ σας παρακαλώ να σημειώσετε ότι συμφωνώ και πρέπει απλώς να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών ομάδων για να καταρτιστεί το, η επιστολή αυτή εγκαίρως. Τώρα ερχόμαστε στο σημείο 20 και Κυρίες και κύριοι, προχωράμε και πρέπει κάπως να επιταχύνουμε. Σχετικά με το επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως, δηλαδή την παρουσίαση της ενδιάμεσης αξιολόγησης της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης καταμερισμού των κινδύνων. Ε, ε, καλωσορίζω την Έρικα Μαν, πρώην συνάδελφό μας και τον Λουκ Σούτε. Ε, ελπίζω ότι όλα είναι σαφή και η κυρία Μαν μπορεί να ξεκινήσει. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μας να βλέπουμε ένα γνωστό πρόσωπο και δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα και εγώ χαίρομαι. Χαίρομαι που βλέπω τόσους συναδέλφους τους οποίους γνωρίζω καλά. Ε, ε, είναι, κάτι καλό. Θα μιλήσω αγγλικά αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα διότι όλα τα έγγραφα που θα δείτε μπροστά σας είναι αγγλικά. Θα πρέπει να έχουν κατανεμηθεί και ε, γι' αυτό θα μιλήσω αγγλικά, θα είναι πιο εύκολο για σας. Αυτό λοιπόν θα σας παρουσιάσω είναι το RSFF, Risk Sharing Finance Facility, κάτι το οποίο ε, στήριξε το Κοινοβούλιο με ένα δισεκατομμύριο σε δύο δόσεις. Στο τέλος λοιπόν του, ε, προτού ληφθεί η απόφαση για το πρόγραμμα πλαίσιο 7 είχαμε ζητήσει στα μέσα της διαδρομής να υπάρξει μία αξιολόγηση και αυτό κάναμε. Τώρα θα συζητήσουμε αυτή την αξιολόγηση. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν να πάρετε την πρώτη διαφάνεια. Όταν κοιτάξετε την πρώτη διαφάνεια... Um, προσπαθήσουμε να δούμε τη δυνατότητα συνεργασίας καθώς και την ε, αξιολόγηση που έλαβε ε, χώρα το 2010. Έγινε μία αξιολόγηση από ανεξάρτητους ε, εμπειρογνώμονες. Επειδή δεν έχουμε τόσο χρόνο, θα ήθελα να δούμε την εμβέλεια του εγχειρήματο γιατί σας ενδιαφέρει άμεσα. Αρχίσαμε φέτος, ήμασταν έξι εμπειρογνώμονες και ξεκινήσαμε. Ο εισηγητής ήταν ο κύριος Σίτε, καθηγητής στο Μάστριχ και ε, επίσης πρίτανης σε ένα από τα πανεπιστήμια του Μάστριχτ. Άρα είχαμε ένα ιδιαίτερα αξιόλογο ε, staff εμπειρογνωμόνων. Η αξιολόγηση έληξε έγκαιρα και είδαμε τα βασικά ζητήματα που έπρεπε να μας απασχολήσουν, δηλαδή να δούμε αυτό το μέσο χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, να δούμε κατά πόσο ήταν συνεκτικό, αποδοτικό, αηφόρο και να δούμε και τις μακροχρόνιες επιπτώσεις. Όταν, ας δούμε, σας παρακαλώ την επόμενη διαφάνεια. Όταν δείτε το μέσον αυτό, νομίζω ότι αυτό που προσπαθήσαμε με αυτό το μέσο ήταν να καλύψουμε τον τομέα της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας. Δηλαδή μιλάμε για την ατζέντα καινοτομίας. Επίσης προσπαθούμε να δούμε τι κάνει και η ΕΤΕ και πώς μπορούμε να προβούμε σε επενδύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το έχουμε ε, ρυθμίσει τα τελευταία χρόνια έτσι ώστε να σταθούμε σε αυτό τον τομέα και να δούμε πώς μπορούμε να διευρύνουμε το πρόγραμμα. Το τρίτο θέμα είναι ότι πρόκειται για μια συγχώνευση μέσων, δηλαδή βασιζόμαστε σε, αυτό το κέριο ζήτημα. Είναι ένα μακροχρόνιο μέσον και τα χρήματα προέρχονται από την αγορά. Η ΕΤΕ διαχειρίζεται τα κονδύλια με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επίτροπης, αλλά τα χρήματα που προήλθαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή ένα εκατομμύρια η πρώτη δόση, η πρώτη δόση 500.000 και άλλες 500.000 αργότερα, θα πρέπει να ε, επιμεριστούν και θα λάβουμε και ένα δις επιπροσθέτως από την ΕΤΕ. Και πρόκειται για ένα κεφάλαιο εγγύησης αν δεν χρησιμοποιηθεί. Είναι κάτι το πολύ σημαντικό, αλλά αυτό το ένα δις, αυτό το, το μαξιλαράκι, αυτό το κεφάλαιο επιτρέπει στην ΕΤΕ να φτάσει σε 10 εκατομμύρια, δηλαδή να βρει από την αγορά 10, 10 ε, δισεκατομμύρια, με συγχωρείτε. Δηλαδή βασιζόμαστε στην έννοια της δανειοδότησης, γι' αυτό είναι ένα από τα καλύτερα μέσα που αναπτύξαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι ομάδες στόχου είναι οι δημόσιοι φορείς, ε, οι ιδιωτικέ επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, οτιδήποτε. Και θα το δούμε αυτό αργότερα, εάν το επιθυμείτε. Αν δείτε την ε, επόμενη διαφάνεια, θα δείτε μία ανακεφαλαίωση για να δείτε την κατανομή των κεφαλαίων, ας λάβετε υπόψη ότι πρόκειται για το τέλος του, μέχρι το τέλος του 2009. Έχουμε και περαιτέρω εξελίξεις. Βλέπετε όμως την κατανομή, δηλαδή τα χρήματα πώς επιμερίζονται, πόσα έχουν εγκριθεί και βλέπετε ότι τα εγκεκριμένα κονδύλια είναι η μεγαλύτερη ε, στήλη. Και αυτά που έχουν εκταμιευθεί είναι η μικρότερη ε, στήλη. Όταν έχετε χρόνο στα γραφεία σας, δείτε αυτή την ανελικτική πορεία, γιατί αρχίσαμε το 2007, αργή ήταν η πορεία το 2008, μετά βλέπετε την ηλικιώδη ανάπτυξη και δύο είναι οι λόγοι γι' αυτό. Καταρχήν η χρηματοοικονομική κρίση ήταν ένα εξαιρετικό μέσο. Ήταν σαν ένα μάνα εξ ουρανού γιατί δεν ξέραμε τι θα συμβεί αρχικά. Είναι ένα από τα λίγα ε, μέσα που λειτουργήσαν στην αγορά και επειδή είχαμε αυτό το εγγυητικό κεφάλαιο μπορέσαμε, μπορέσαμε να εκταμιεύσουμε χρήματα από την αγορά διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να εκταμιευθούν τόσα χρήματα αν δεν υπήρχε αυτή η κεφαλαιοχική εγγύηση. Άρα αυτό το στοιχείο θα επαυξηθεί και στο μέλλον. Επίσης, θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι βρισκόμαστε πέραν από τα αρχικά προβλεπόμενα στοιχεία. Είμαστε στο 5,5 δις τώρα. Τα στοιχεία που βλέπετε ανέρχονται στο, στα 6 δις. Και τώρα, το 2010, είμαστε πολύ κοντά στα 8 δις. Θα ήθελα να αναφερθώ στον John David Marlowe και την ομάδα του που μας βοήθησαν και τον Μακ Τόγκερ από την ε, ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δείτε την ε, ανωδική πορεία λοιπόν και λάβετε τη σοβαρά υπόψη. Αν δείτε την επόμενη διαφάνεια είναι πολύ ενδιαφέρουσα διότι σας δίνει μία ανακεφαλαίωση για το τι μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Βλέπετε ότι τα όλα μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Ε, γίνεται μία έρευνα για ένα πρόγραμμα οικονομικής καθαρά εφαρμογής. Γι' αυτό που μας ενδιαφέρει αν το σημείο κίνησης είναι καλό για να φτάσουμε σε προϊόντα νέας γενεάς. Άρα περνάμε από φάση πανεπιστημιακή, καθαρά πανεπιστημιακής έρευνας σε επιχειρηματική εφαρμογή. Αν δούμε την επόμενη διαφάνεια, εδώ έχετε μια συνολική εικόνα για την ταξινόμηση των σχεδίων RSFF, δηλαδή ως προς το χρηματοδοτικό μέσο καταμερισμού των κινδύνων, πώς ανελήχθηκε το... Τώρα βρισκόμαστε σε φάση 7 προγραμμάτων. Δεν, δεν θα ήθελα να σας απασχολήσω περισσότερο, διότι θα χρειαστεί πολύς χρόνος. Εδώ στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε κάτι πολύ ενδιαφέρον, γιατί βλέπετε ε, τη συμμετοχή από τα, των κρατών μελών και των συνδεδεμένων κρατών. 19 κράτη-μέλη και δύο συνδεδεμένες χώρες συμμετέχουν. Το Μεγαλύτερο μερίδιο είναι αυτό της Γερμανίας. Υπάρχει ένα αριθμητικό στοιχείο που θα, θα, θα σας εκπλήξει. Βλέπουμε πολύ, ότι είναι πολύ χαμηλή η συμμετοχή της Γαλλίας, 6,4. Αυτό ισχύει γιατί η Γαλλία έχει ένα παράλληλα ε, εθνικό πρόγραμμα. Γι' αυτό μπορεί να ερμηνευτεί αυτή η χαμηλή ποσοστή αναλογία. Από την άλλη πλευρά βλέπετε από τα νέα κράτη-μέλη στοιχεία. Η Ουγγαρία πολύ υψηλή συμμετοχή, Πολωνία, συνδεδεμένες χώρες ε, στην έρευνα και ανάπτυξη συμμετέχουν κατά πολύ η Ισραήλ, Τουρκία. Το Ισραήλ είναι υπαριθμόν ένα χώρα και θα κατανοήσετε από την επόμενη διαφάνεια γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο. Διότι σχετίζεται με έναν από τους τομείς έρευνας. Έχετε λοιπόν μία συνολική εικόνα ως προς την κατανομή ανατομέα. Δεν μας εκπλήσει καθόλου όμως είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να το δούμε, διότι στην έρευνα στο τομέα της μηχανικής, η έρευνα στο τομέα της μηχανικής έχει το μεγαλύτερο ε, μερίδιο και βλέπουμε ότι στη Life Science έχουμε μεγάλη αύξηση ανά την Ευρώπη και εδώ βλέπουμε ότι το Ισραήλ συμμετέχει ενεργά. Γιατί συμβαίνει αυτό. Θα σας το αναπτύξω κάποια μέρα. Ίσως θα μπορούσατε να καλέσετε κάποιον από το Ισραήλ κάποια μέρα από το Υπουργείο Έρευνας, διότι το Ισραήλ επενδύει σε αυτό το τομέα με διαχείριση ε, από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στον τομέα της ενέργειας και το τομέα ICT, δηλαδή καινοτομία, επικοινωνία και τηλεπικοινωνίες. Εδώ υπάρχει ε, μεγάλη συμμετοχή από όλους. Θα το δούμε αργότερα. Ως προς το, ε, το θέμα του επιμερισμού συζητήθηκε και με τον Γενικό Διευθυντή, τον κύριο ε, Γιάν Σμίτς. Θα ήθελα η Επιτροπή και η ΕΤΕ να μας μιλήσουν περισσότερο. Φαίνεται απλό, αλλά είναι πολύ περίπλοκο να φτάσετε σε αυτά τα αριθμητικά στοιχεία. Βλέπετε ένα 60% που αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις. Όταν μιλάμε για μεγάλες επιχειρήσεις, σημαίνει ότι λαμβάνουν τα χρήματα. Έτσι ίσως εννοείται, όμως όταν δείτε το πρόγραμμα δεν σημαίνει ότι μια μεγάλη επιχειρήση έρχεται και παίρνει τα χρήματα, θέλει δηλαδή ένα δάνειο από την αγορά. Πρόκειται για ένα συγκεκριμένο σχέδιο που σχετίζεται με κάτι το ιδιαίτερο γιατί μην ξεχνάτε ότι πάντα πρέπει να καλύπτουμε αυτό το, το στοιχείο κινδύνου. Άρα δεν μπορεί να διασπαθιστεί το χρήμα από επιχειρήσεις. Ακόμα λοιπόν και για την Κρούπς ή και για την Φίλιπς, γιατί εδώ έχουμε ε, ένα σχέδιο καινοτομίας που προωθεί η Φίλιπ στο Eindhoven ε, καλύπτει ένα κλάστερ, μία ομάδα ΜΜΕ. Δηλαδή 40 ΜΜΕ, περισσότερο δηλαδή, περισσότερες από αυτές που αναφέρονται εδώ, προέρχονται από όλη την Ευρώπη και από άλλες χώρες και ομαδοποιούνται σε ένα μεγάλο ε, project στην, στο Eindhoven. Μπορείτε δηλαδή να το δείτε αυτό το συγκρότημα από τον αυτοκινητόδρομο. Αυτό να λαμβάνετε υπόψη όταν βλέπετε ένα 60%. Το ίδιο αφορά τις ΜΜΕ και τα, το, τους, ε, τα ανώτατα όρια. Μπορώ να σας δώσω στοιχεία για τις ΜΜΕ μέχρι το τέλος του 2009 είχαμε δύο ΜΜΕ, τώρα έχουμε ε, λίγο περισσότερες το 2010 που την χάνουν αξιολόγησης, αλλά σε, αυτό, σε αυτή την ομάδα ε, επιχειρήσεων έχουμε το μέτενβες το Eindhoven, και υπάρχουν και πολλές ΜΜΕ στο παρασκήνιο. Γιατί υπάρχει μία πλατφόρμα που ε, βοηθά τις ε, ΜΜΕ. Ως προς τα mid-caps κάναμε μία αποτίμηση και φτάνουμε στους χιλίους υπαλλήλους, από χιλίους υπαλλήλους τις, στους 2.000 δηλαδή. Μιλάμε για τις κλασικού τύπου ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και βλέπετε ως προς τα πανεπιστήμια καλύπτονται και αυτά και θα ήθελα να δείτε το Πανεπιστήμιο Κολίνσκα από τη Σουηδία Εξαιρετικό είναι αυτό το πρόγραμμα, το κλινικό του σκέλος, στο κλινικό του σκέλος. Και θα ήθελα από τη δική σας πλευρά ως μέλη του Κοινοβουλίου να το δείτε αυτό, διότι σε ορισμένα κράτη-μέλη όπως τη Γερμανία τα πανεπιστήμια δεν μπορούν να χρησιμοποιούν αυτού του τύπου δάνεια. Δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο δια νόμου. Θα ήθελα να το δείτε, διότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα προσκόμματα και δεν έχει νόημα. Γιατί τα πανεπιστήμια τη στιγμή που ε, προωθούν, δημιουργούν εισόδημα, ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας, δεν έχει νόημα να μην μπορούν να χρησιμοποιούν δάνεια. Δείτε μόνο έναν αριθμό εδώ, σε αυτή τη διαφάνεια, είναι η συνολική επένδυση. Θα ήθελα να σας πω ότι το ένα δις προέρχεται από τον προεχειρισμό, φτάνουμε στα 10 δις από την αγορά και μετά έχουμε άλλα 6 δις που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό είναι εξαιρετικό εκθαμβωτικό αυτό το μέσον, διότι τα χρήματα που μπορούν να διατεθούν είναι πάρα πολλά. Τώρα, ως προς τα συμπεράσματα, εντάχει, όπως σας είπα και πριν, μας ενδιαφέρει ο καινοτόμος χαρακτήρας, η κατά περίπτωση αποτίμηση που μπορεί να αλλάξει διαχρονικά. Γιατί από τότε που γνωρίσαμε τη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση ήταν δύσκολο να μπορέσουμε να προωθήσουμε τέτοιες δανειοδοτήσεις. Αυτό το σχέδιο ήταν το μόνο, αυτό το ε, σχήμα ήταν το μόνο που ήταν διαθέσιμο στην αγορά. Θα ήθελα λοιπόν να μην σταματήσουμε αυτή τη διαδικασία μετά από τη λήξη του εβδόμου προγράμματος πλαισίου, αλλά να το προωθήσουμε ε, περαιτέρω. Πρόκειται λοιπόν για ένα πολύ ενδιαφέρον μέσον. Υπάρχουν δέκα συστάσεις ε, στη συνέχεια, οι οποίες είναι οι εξής τις έχουμε ομαδοποιήσει σε δύο περιόδους. Η πρώτη είναι το 2011 έως 2013, αυτή είναι η πρώτη χρονική περίοδος και το πιο σημαντικό είναι ότι χρειαζόμαστε τη δική σας υποστήριξη. Βλέπω ότι ο Κρίστιαν Ήλερ και πολλά μέλη μας βοήθησαν ιδιαίτερα στο, ε, στη δημιουργία αυτού του προγράμματος γι' αυτό. Θα πρέπει να έχουμε 500 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη συνεργασία και από τον τομέα των δυνατοτήτων. Αυτό ήταν μέρος της ε, συμφωνίας και της νομικής βάσης για το πρόγραμμα πλαίσιο το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. 400 δηλαδή εκατομμύρια από τη συνεργασία και 100 από, τις, ε, από το τομέα των ε, ικανοτήτων. Αυτό γνωρίζω ότι μπορεί να θέσει ορισμένα επιμέρους προβλήματα, αλλά θα θέλαμε να μας υποστηρίξετε. Θα πρέπει να έχετε κατά νου ότι βρισκόμαστε πέραν από το δίκτυ που αναμέναμε. Βρισκόμαστε στα 8 δις εγκεκριμένων κονδυλίων, δηλαδή χρειαζόμαστε 2 δις, απομένουν 2 δις μέχρι το 2011, άρα οι προσδοκίες της ΕΤΕ είναι ότι μέχρι την άνοιξη καλοκαίρι, αν δεν έχουμε τα 500 εκατομμύρια θα πρέπει να κλείσουμε το πρόγραμμα το οποίο θα ήταν ε, κρίμα πραγματικά διότι η κρίση δεν έχει ε, λήξει και τα καινοτόμα σχέδια θα πρέπει να, προ... να προωθηθούν. Τα προγράμματα αυτά υπάρχουν και θα ήταν κρίμα να σταματήσουν εδώ. Ξέρω ότι ε, είναι μεγάλο το άχθος των, ε, των ετοιμάτων μας, αλλά μιλάμε για 500 εκατομμύρια και το αφήνουμε σε εσά να δείτε ποιοι πόροι, πόσοι πόροι είναι διαθέσιμοι, διότι ακόμα και αν εκταμιευθούν τα 500 εκατομμύρια, δεν θα είχαμε επαρκείς εγγυήσει μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. Γι' αυτό είμαστε πολύ κοντά και θα ήταν κρίμα εάν δεν θα μπορούσε αυτό το μέσο χρηματοδοτικής διευκόλυνσης να μην είναι λειτουργικό μετά το 2011. Χρειαζόμαστε τα 500 εκατομμύρια, τα επιπρόσθετα 500 εκατομμύρια γιατί εμείς ήμασταν σε θέση να φτάσουμε σε 5 ε, δις αρχικά και αυτό ήταν το πρότυπό μας. Μετά το 2013, εντάχει να σας πω, ότι η σύστασή μας έχει ως εξής. Αν δείτε πόσα, σε τι ε, υψηλά ποσά φτάσαμε από τις μεγάλες επιχειρήσεις, από τα πανεπιστήμια και ούτω καθεξής, θα θέλαμε να αυξήσουμε το, την κεφαλαιοχική βάση σε 5 δις. Αυτό δεν θα χαθεί. Θα ε, χρησιμοποιηθεί μόνο αν υπάρχει αποτυχία κάποιου σχεδίου, το οποίο μπορεί να ε, επισυμβεί. Διαφορετικά τα χρήματα θα παραμείνουν και θα αυξηθεί και ο τόκος. Ήταν ένα ιδιαίτερα ευφυές μέσον. Φτάσαμε σε εκταμίευση χρημάτων από την αγορά και φτάσαμε στο 1,5 δις. Αλλά αυτό θα πρέπει να σας απασχολήσει όποτε θέλετε περισσότερες πληροφορίες πληροφορίες. Η Επιτροπή και η ΕΤΕ θα μπορέσουν να σας δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και πολύ, με πολύ ε, ε, γρήγορους ε, ρυθμούς. Άρα μετά από δυόμιση χρόνια ίσως δεν θα πρέπει να γίνει η κλασική αξιολόγηση αλλά μία άλλη αποτίμηση με ένα μεγαλύτερο δίκτυο ασφαλείας. Για να μην υπάρχουν επικαλύψεις επίσης στα χρηματοοικονομικά σχέδια. Εδώ χρειάζεστε λίγο χρόνο. Η ΕΤΕ ε, ε, κάνει λόγο για κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου. Εδώ γνωρίσαμε μεγάλη επιτυχία. Αλλά πολλές φορές μπορεί να υπάρχει επικάλυψη. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς έχουν να αποτιμήσουμε όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα και να δούμε τι προβλέπεται και για ποιο σκοπό. Για ποιο σκοπό. Αυτό όμως αποτελεί μια δική μας σύσταση. Υπάρχουν ε, ορισμένα ερωτήματα τα οποία θα ήθελα να δούμε μαζί. θα πρέπει να δούμε κατά πόσο έχουμε ορίσει τους στόχους και κατά πόσο έχουν εφαρμοστεί Δηλαδή, με βάση το σχέδιο. Ναι, πολύ αποτελεσματικά. Είχαμε μια εξαιρετική ομάδα στην ΕΤΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να συνεχίσει αυτή η ομάδα το έργο της που ήταν ιδιαίτερα επιτυχές. Ποια ήταν τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες. Ήταν ένα αντικυκλικό μέσο κατά τη διάρκεια της κρίσης έχει ένα μεγάλο περιθώριο μόχλευσης, μπορεί να εκταμιεύσει χρήματα από την αγορά, είναι πολύ αποτελεσματικό στην εφαρμογή του. Τώρα, οι ε, αδυναμίες είναι η υποδομή των ΜΜΕ, αλλά εν πάση περιπτώσει όχι τόσο όσο ε, νομίζαμε στην αρχή. Θα δούμε, και αν δούμε τις λεπτομέρειες, μπορούμε να είμαστε κάπως ήσυχοι. Ως προς υποδομές αποτελούν ένα μεγάλο πρόβλημα. Θα ήταν σκόπιμο να έχουμε περισσότερα σχέδια υποδομών για να εφαρμοστούν με βάση αυτό το μέσον. Και θα ήθελα να σας πω κάτι ε, κάπως ε, εξαπίνηση είναι το ευρωπαίνα Ξέρω ότι σας ενδιαφέρει αυτό το μέσο, το οποίο ίσως να είναι οι ιδεώδες. Δεν έχει αποτιμηθεί ακόμα. Βασιζόμαστε στη ζήτηση, υψηλή ζήτηση, δηλαδή όταν, υπάρχει, όταν υπάρχουν υπερβολικές ε, εγγραφές, δηλαδή πολύ υψηλότερες από το αναμενόμενο, αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό. Ποια είναι τα αποδεικτικά στοιχεία, τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Έχουμε την ε, σημαντική γεωγραφική κάλυψη, έχουμε μια μεγάλη γεωγραφική κάλυψη και ορισμένες, ορισμένα, ορισμένες ε. συμμετέχουν αρκετά. Τι μπορούμε να βελτιώσουμε τώρα. Σας προτείνουμε να να δούμε γιατί δεν μπορούμε να δελειάσουμε τις ΜΜΕ ενώ καλύπτονται αρχικά. Θα πρέπει να καταβάλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες και ο εισηγητής μας έχει απαντήσεις. Ασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Ένα άλλο θέμα που απασχόλησε την ΕΤΕ είναι να έχουμε εταίρους στα κράτη-μέλη. Αν δεν κάνω ε, λάθος έχουμε μόνο δύο εταίρους. Αυτό τι σημαίνει. Θα θέλαμε να έχουμε σαφείς ενδείξεις από ε, εταίρους όπως η ΕΤΕ ή άλλους εταίρους που θα συνεργαστούν με την ΕΤΕ είναι πώς μπορούμε να διανοίξουμε ένα δρόμο για τις ΜΜΕ και να αντισταθμίσουμε το, το μέρισμα κινδύνου, την συνιστόσα μάλλον του κινδύνου και από πλευράς κράτους μέλους για να μπορέσουμε να εκταμιεύσουμε ακόμα περισσότερα χρήματα από την αγορά και να έχουμε ΜΜΕ από την Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Ουγγαρία και ούτω καθεξής. Ε, λειτουργεί πάντως πολύ καλά κάτω από το 5,5, κάτω από το 7,5 ε, εκατομμύρια θα πρέπει να εκτελεστεί το project από το κράτος μέλος. Θα θέλαμε να δείτε και ορισμένα άλλα στοιχεία όπως ε, το equity funding και να δείτε ποιες είναι οι μελλοντικές προοπτικές που διανοίγονται. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο έγγραφο και θα συγκεράσουμε όλες αυτές τις ιδέες από κοινού. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ για αυτήν την πολύ λεπτομερή ε, παρουσίαση και ο πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Έλε. Ευχαριστώ, θέλω να σας ευχαριστήσω. Είμαι ο τελευταίος που επιβίωση του τριμερούς διαλόγου. Είχαμε τότε κάνει τρεις ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή, 30 ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν μπόρεσα να απαντήσω σε μία. Και πρέπει να σας πω ότι έχω διαβάσει πάρα πολύ ε, προσεκτικά ε, το κείμενο και η έκθεση ουσιαστικά ε, αναφέρεται σε διάφορα από τα ερωτήματα που είχαμε θέσει τότε τότε είχαμε πει ουσιαστικά ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έπρεπε να δίνει περισσότερα αλλά έπρεπε να υπάρχουν και περισσότερες εθνικές παρεμβολές διότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ήθελε να κρατήσει πολύ μεγάλες τις δόσεις και εμείς θέλα, η πιο μικρή ε, δόση ε, θέλαμε να είναι ε, 5 εκατομμύρια διότι ε, για κάθε μεγάλη δόση η Τράπεζα Επενδύσεων και κερδίζει πολλά χρήματα και δεν έχει πολλή δουλειά. Ε, ε, έπρεπε λοιπόν να υπάρχουν εθνικοί μεσάζοντες και μία ανισομερής κατανομή μέσα στη χώρα. Πράγμα το οποίο δεν είναι πολύ προφανές και ίσως οφείλεται στο ότι υπάρχουν μεσάζοντες, δεν υπάρχουν μεσάζοντες εθνικοί σε μικρότερες χώρες όπως η Ρουμανία και είναι δύσκολο σε τέτοιες χώρες να αναλάβουν τόσο μεγάλα δάνεια. Όσον αφορά την τάξη μεγέθους των δόσεων όπως ανέφερα, εάν θέλουμε να έχουμε περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να ε, μειώσουμε το μέγεθος των δόσεων διότι ε, μία μικρομεσαία επιχείρηση με μάξιμουμ 250 απασχολούμενους ε, δεν μπορεί να αφομοιώσει 5 εκατομμύρια άρα θα πρέπει να μειώσουμε το μέγεθος των δόσεων άρα το καθεστώς αυτό γίνεται πιο δαπανηρό ή θα πρέπει πρέπει να έχουμε μία ρύθμιση ευρωπαϊκού επίπεδου οπότε θα μπορούσαμε να παραμείνουμε στις δόσεις αυτές και να τις ρυθμίσουμε εσωτερικά. Είναι θέμα ε, πολιτικής απόφασης. Ένα άλλο θέμα Ε, το οποίο ε, ε, έθεσα και έθεσε προηγουμένως ο κύριος Κούντς. Είχαμε πει 500 εκατομμύρια στην αρχή και μετά θέλαμε να πάρουμε από το πρόγραμμα ακόμη 500 εκατομμύρια. Αλλά πρέπει να δούμε και το κόστος σκοπιμότητος. Δηλαδή υπάρχει μαζί με τη μόχλευση μία, ένα προσόν στο να καλύψουμε αυτά τα δισεκατομμύρια και μετά θα πρέπει να αφαιρέσουμε από το πρόγραμμα ένα δισεκατομμύριο. Άρα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα η Επίτροπος να μας δώσει μία πολιτική απάντηση διότι ε, αν θέλουμε να προωθήσουμε την ανάπτυξη και την καινοτομία να μην μας λέει ότι αυτά έχουν χρηματοδοτηθεί για να υπάρξει ε, έρευνα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό η Επίτροπος να το θέσει σε ένα γενικότερο πλαίσιο, να διαχωρίσουμε δηλαδή ποιο ε, ποσοστό ε, θα αποδοθεί στην καινοτομία και ποιο στην κλασική έρευνα. Επίσης, καλό θα ήταν να μελετήσουμε και να επαληθεύσουμε ε, ποιοι είναι οι πραγματικοί παράγοντες καινοτομίες. Γιατί αν μιλάμε δηλαδή για μια επιχείρηση επιχείρηση σαν την Philips στις ε, ε, ε, ε, στις μεγάλες επιχειρήσεις ο τομέας καινοτομίας χρηματοδοτείται εσωτερικά κατά 11-12% δηλαδή ένα ποσοστό 11-12-15% του ποσού αντλείται μέσα από την επιχείρηση με ένα τέτοιο λοιπόν εργαλείο θα είχαμε τη δυνατότητα να, να μην αναφερθούμε καν στην καινοτομία διότι το εσωτερικό ο κόστος της ε, καινοτομίας θα εξωτερικευτεί ε, και ε, μπορεί ίσως να υπάρξουν πιο ενδιαφέροντες αναχρηματοδοτήσεις προγραμμάτων. Δεν θέλω να, να απαντήσω τώρα αλλά είναι ένα ερώτημα που πρέπει να θέσουμε, διότι κατά τη διάρκεια της κρίσεως ε, υπήρχε κάποιος λόγος για τον οποίο χρησιμοποιήσαμε αυτό το μέσο με αυτόν τον τρόπο, διότι μειώθηκαν ε, τα ποσοστά καινοτομία για να μπορέσουν να δανειστούν στις κεφαλαιαγορές οι επιχειρήσεις. Όταν όμως θα υπάρχει μια φυσιολογική κατάσταση ε, θα μπορούσε να εξεταστεί εάν ε, η εσωτερική χρηματοδότηση κατά κάποιον τρόπο επιδότηση είναι σκοπιμότερη ή πρέπει να υπάρξει εξωτερική χρηματοδότηση για την καινοτομία κατά τρόπον ώστε να ε, βρούμε μεθόδους να χρησιμοποιήσουμε μεγάλα κεφάλαια και ε, βέβαια η τράπεζα έχει συμφέρον να δίνει μεγάλες πιστώσεις για να κερδίζει πολλά χρήματα. Άρα, ερώτηση, πώς θα υπάρξει προτιθέμενη αξία σε αυτό τα δάνεια για την Ευρώπη, διότι τότε είχαμε ε, ρωτήσει και υπήρχε μία πολύ σαφή εικόνα και εφόσον τώρα έχουμε ένα μέσο που λειτουργεί ομαλά, μπορούμε να πούμε ότι, δεν, ε, ε, ε, ότι θα διαθέσουμε τα 500 επόμενα εκατομμύρια, αλλά μόνο εφόσον ξέρουμε ποιες είναι οι προοπτικές και οι προϋποθέσεις του προϋπολογισμού. Διότι εδώ πήραμε ένα δισεκατομμύριο από την έρευνα και το τροφοδοτήσαμε την καινοτομία της βιομηχανίας αλλά αυτό δεν πρέπει να αποτελέσει την κατεύθυνση για το μέλλον διότι θα ε, ε, ε, μειώνουμε συνέχεια το ερευνητικό μας προϋπολογισμό προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει να υπάρξουν νέοι πόροι και όχι μείωση των ε, κλασικών πόρων για ε, την έρευνα. λοιπόν. ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Η επιτυχία ε, πέρα του, του εγχειρήματο. όπως ερμηνεύεται εδώ πέρα από την Έρικα Μάν, όχι μόνο ως πρόεδρος της Επιτροπής ε, Αξιολόγησης. Νομίζω πως ε, έχει εδώ πέρα λειτουργήσει. Δηλαδή έχουμε ένα μέσο το οποίο είναι τελείως καινούριο και υπήρχαν πάρα πολλές αντιρρήσεις για να πάρουμε λεφτά από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και να πάνε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και πρέπει να το κρίνουμε ως εξής να δούμε πως η μόχλευση ε, έχει έναν ε, πάρα πολύ υψηλό βαθμό ολεκλήρωση. Εγώ είχα την ιδέα πως ε, θα ενισχύαμε τις ε, υποδομές και βλέπουμε εδώ πέρα πως παρότι ότι μεταφέρονται πάρα πολλά λεφτά από εκεί πέρα παραμένουν ε, εκτός ή τέλος πάντων παραμιλημένες οι υποδομές κάτι το οποίο μου προξενεί εντύπωση κατόπιν ναι και εγώ ε, συμφωνώ με το ερώτημα το οποίο μόλις ε, ακούστηκε για τις μεγάλες ε, εταιρείε οι οποίες θα πρέπει να αναχρηματοδοτήσουν για να κάνουν αυτά τα, τα πράγματα οπότε πραγματικά τι είναι εδώ πέρα η προσθέμενη αξία που δεν μπορούσε να επιτευχθεί αλλιώς και τέλος είμαι θετικός, ε, δεν ξέρω, στο να κοιτάξουμε τα, τα διαρθρωτικά ταμεία. Δεν είναι ανάγκη όλα αυτά να προέλθουν οπωσδήποτε από τη μεριά της έρευνας. Εντάξει, βεβαίω ε, όταν μιλάμε για την καινοτομία υπάρχει νομίζω μια σελίδα που είναι τα, τα 10 αυτά σημεία. Θα δείτε εκεί πέρα κάτω στην ε, καινοτομία να έχουμε ένα δισεκατομμύριο από τα διαρθρωτικά ταμεία να σκεφτούμε ίσως πιο δημιουργικά και όχι μόνο στην σημερινή περίοδο. Αυτά. Ευχαριστώ. Η Αγγέλικα Νίμπλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω για το ότι η αγαπητή συνάρφος επί σειρά ετών η κυρία Μαν είναι ξανά εδώ πέρα στο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ειδικό και να πω πως αποτελεί μια εγγύηση ποιότητας ε, και χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Έχω και εγώ ένα ερώτημα που ανέφεραν και οι δύο προλαλήσαντες στις ε, γραπτές εξηγήσει εδώ πέρα αναφέρετε σαφώς πως δεν μπορέσατε να έρθετε σε επαφή με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οπότε δεν ξέρω, αυτό γίνεται μέσω ενδιαμέσων, μέσω των κρατών μελών, ίσως έτσι θα μπορούσαμε να υπάρξει μια οικονομική στήριξη μέσω των τραπεζών επιτόπου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μου φαίνεται λογικό αυτό και μια καλή προσέγγιση. Και οι ειδικοί το ίδιο πριν Και μετά να αναφέρω κάτι το οποίο με εξέπληξε και θα ανέφερε και ο κύριος Φανίστελ Ρόι, πως για την ερευνητική υποδομή δεν χρησιμοποιήθηκε αυτό το μέσο σχεδόν καθόλου. Και εγώ περίμενα κάτι ε, διαφορετικό γιατί συζητάμε εδώ πως θα πρέπει να εκδώσουμε ευρωομόλογα δεν χρηματοδοτούμε δηλαδή μόνο τα ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα αλλά και την, τις υποδομές της ενέργειας οπότε νομίζω πως αυτό το μέσο θα ήταν ιδιαίτερα ενδεδειγμένο για να χρησιμοποιηθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το ερώτημα μου είναι, έχετε κάποια εξήγηση για το γιατί το RSFF ε, χρησιμοποιήθηκε τόσο λίγο σε αυτό το τομέα. Και τέλος, τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά έτσι ώστε το μέσο αυτό, το οποίο θα έπρεπε να είναι νομίζω οπωσδήποτε αποδεκτό, να γίνει ακόμη πιο ελκυστικό. κυρία Ριέρα Μαδρουέλη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Μαν, είναι μεγάλη μας ευχαρίστηση να σε έχουμε εδώ απόψε και συγχαρητήρια σε όλους σας για την καλή δουλειά που έχετε κάνει. Σε με τον κύριο Έλτερ, εγώ δεν εκπλήσω, γνωρίζομαι πως υπάρχουν κάποιοι λαμπροί άνθρωποι σαν και σας ε, στις τάξεις των σοσιαλιστών, όχι μόνο στον τομέα της οικονομίας αλλά και σε άλλους ε, τομείς. Συμφωνώ μαζί σας όταν λέτε πως το RSF είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μέσο το οποίο ε, έχει λειτουργήσει αρκετά καλά και θα πρέπει να συνεχιστεί με το πρόγραμμα πλαίσιο 7 και εμείς ε, είχαμε την εντύπωση πως λειτουργεί καλά για ορισμένα έργα, ειδικά τα μεγάλα βιομηχανικά έργα ή τουλάχιστον έργα κάποιου μεγέθους και πάνω, αλλά ίσως να μην ε, λειτουργεί τόσο καλά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εσείς μιλήσετε για συγκεκριμένα παραδείγματα ομάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που περιλαμβάνουν και κάποιε μεγάλε εταιρείε και σε αυτέ τι περιπτώσει πράγματι λειτουργεί, αλλά δεν λειτουργεί καλά με ομάδε ερευνητών που ίσως να ασχολούνται με πιο ρηψοκίνδυνα έργα, τα οποία όμως είναι οπωσδήποτε ποιοτικά. Επίσης, ε, κάνατε λόγο για τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά εγώ θα ήθελα να γνωρίζω τι σκέφτεστε για το πώς θα μπορέσουμε να τις συμπεριλάβουμε. Τώρα θα δώσω τον λόγο στην κυρία Μαν και στον κύριο Σουτ για να απαντήσουν. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Θα είμαι πολύ σύντομη και μετά ο, ο κύριος Σούτ θα κάνει την, το επόμενο τμήμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που πιστεύετε ότι είναι ε, καλός ο τρόπος με τον οποίο κάναμε την παρουσίαση. Όσον αφορά τον συνάδελφο Έλερ, και την Αγγέλικα Λίμπλερ. Δύο θέματα θέλω να θίξω και θα είμαι πολύ προσεκτική. Θα δω ακριβώς τι εννοούμε με ε, τον όρο βιομηχανική καινοτομία, διότι μπορούμε να σας δώσουμε όλες, ε, όλο το υπόβαθρο και να δείτε όλα τα προγράμματα, διότι στο παρελθόν υπήρχε πάντοτε ένα κενό. Δηλαδή, ε, είχαμε ρίξει χρήματα συνέχεια ή στην έρευνα και μετά τελειώνανε τα χρήματα και όσοι ε, ήθελαν να χρηματοδοτηθούν στην αγορά ήταν μόνοι τους και έπρεπε να ψάξουν να βρουν επιστώσεις ενώ υπάρχουν θέματα τα οποία προχωρούν σε επιχειρήσεις, σε πανεπιστήμια και αν δούμε ουσιαστικά το ποσοστό της οικονομικής έρευνας ε, ε, ε, νομίζω ότι βρισκόμαστε στο 50-60% αλλά πρέπει πάντοτε να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τους υπολογισμούς μας αλλά είναι κάτι που θα μπορέσω να σας δείξω στη συνέχεια και τώρα το δεύτερο θέμα είναι το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχουμε δύο αυτούσια προγράμματα τα οποία θα ολοκληρωθούν το 2010 αλλά σε αυτό το κλάστερ της Philips μέτρησα ότι υπάρχουν περίπου 40 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εμπλέκονται. Στο Medinvest νομίζω και σε με άλλη κατηγορία υπάρχουν 5 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που καλύπτονται από αυτές. Είναι λοιπόν κάτι που πρέπει να ξανασυζητήσουμε διότι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται ένα πλαίσιο και αυτό δεν είναι κακό, είναι πολύ πιο υγιές είτε πρόκειται πρόκειται ή για τον τομέα life science ή για την ενέργεια χρειάζονται ε, να ενταχθούν σε ένα χώρο και ενδεχομένως αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω μεσαζόντων ε, ή ε, με σάζουσες τράπεζες ντόπιε της περιοχής οι οποίες μπορούν να ανοίξουν αυτές τις πιστώσεις αλλά είναι πιο δύσκολο. Μην ξεχνάτε λοιπόν Λοιπόν, γιατί αυτό συνέβη την κατάσταση των ε, εθνικών ε, τραπέζων, ε, τραπεζών μέσα ζώντων τα τελευταία χρόνια. Δεν θέλαν να χάσουν την, τον καθορισμό τους σαν βαθμολογία 3α. Οπότε εάν χάναν αυτή τη βαθμολόγησή τους και χρηματοδοτούσαν κάτι το οποίο δεν ήταν σίγουρο ότι θα απέδιδε, ε, η κατάσταση θα ήταν κρίσιμη. <coughs> Μόλις λίγο ε, χαλαρώσει η κατάσταση, φαντάζομαι ότι αυτές οι δυνατότητες θα βελτιωθούν. Και ο κύριος ε, Λουίκ Σέτερ θα αναφερθεί τώρα εις τις υποδομές και στα πανεπιστήμια. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Έλερ και την προηγούμενη παρατήρηση του διότι αυτό είναι το, η μετακίνηση που κάνουμε στο παράδειγμα και είναι δύσκολο να αξιολογήσουμε τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Ε, αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να αξιολογήσουμε κάτι μεσοπρόθεσμα. Οι ενδείξεις λοιπόν που έχουμε για την ε, συμμετοχή των ε, μεγάλων εταιριών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των εταιριών μέσης κεφαλαιοποίησης αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο η αγορά αντιλαμβάνεται την κατάσταση. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, κάναμε ορισμένες συστάσεις και είπαμε ότι τα 7,5 εκατομμύρια ή ήταν πάρα πολύ η ε, ψηλό ποσοστό όπως είπε η Έρικα προηγουμένως και προχωρήσαμε με ε, το ε, όρο frisbee και όπως είπε ο κύριος Βανίστερ Ρόι δεν πρέπει να περιμένουμε στο 2013 για τα διαρθρωτικά ταμεία τα οποία θα μπορούσαν να εμπλακούν πολύ πιο άμεσα με τις μικρές τράπεζες και ε, θα ολοκληρώσω με τις υποδομές που αναφέρονται στο μέλλον. Εδώ έχουμε έλλειψη 250 εκατομμυρίων, αλλά μπορεί να είναι πολλά χρήματα, δεν ήταν όμως αυτό το οποίο αναμέναμε. Υπάρχει μία μετατόπιση σε χρηματοδότηση εις ε, βάθος αλλά η κατανομή του κινδύνου πρέπει να είναι διαφορετική αν έχετε διαφορετικές δομές και ένα ε, συνεχές ε, έσοδο από την ε, υποδομή δηλαδή ορισμένες ασχολούνται με ουσιαστική έρευνα είναι σε θέση να αποπληρώσουν μέρος του δανείου αλλά ίσως όχι με τον τρόπο που έχει προβλέψει και ε, πρέπει να εξετάσουμε και την αρχή της ε, ζημίας, δηλαδή η ίσως ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καλύπτει τη χρηματοδότηση της πρώτης ζημιάς, της πρώτης απώλειας, first loss και ε, δεν ξέρουμε ακριβώς ε, πού βρίσκεται το ποσοστό της συμμετοχής στην ανάληψη κινδύνου σε αυτό το θέμα. Ίσως λοιπόν ορισμένα από αυτά τα μέσα θα πρέπει κάπως να διορθωθούν εάν η αγορά έχει έλλειψη ενδιαφέροντος για τέτοια θέματα. Επίσης ε, στα πανεπιστήμια υπάρχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, είναι ακόμη πιο περίπλοκα, πολλοί δεν επιτρέπουν που στα πανεπιστήμια να αναλάβουν δάνεια και να χρηματοδοτηθούν κατά αυτόν τον τρόπο. Ε, παραδείγματος χάρη ε, βλέπουμε ότι υπάρχει χρηματοδότηση της, ε, των πανεπιστημίων της, της Μεγάλης Βρετανίας που χρηματοδοτούνται από τράπεζες. Βλέπουμε όμως και την Καρολίνσκα όπου και εκεί υπάρχει μια διαφορετική δομή. Όλα αυτά πρέπει ε, να εξεταχθούν Ο κύριος Φόρτ θέλει να προσθέσει κάτι. Αλλά αν αρχίσουν όλοι με ε, επερωτήσεις δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Με συγχωρείτε, αλλά ήμουν σε μια άλλη επιτροπή. Θέλω να κάνω ορισμένες ερωτήσεις γιατί δεν είχα καταλάβει. Στην πρώτη σελίδα είπατε ότι δεν υπάρχουν επιδοτούμενα δάνεια. Αλλά είτε υπάρχει αγορά, είτε κανείς δεν αναλαμβάνει τον κίνδυνο σε αυτή την τιμή. Είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει. Ε, ε, για μένα σαν, σαν χρηματοδότη αυτό δεν μου φαίνεται ε, πάρα πολύ λογικό διότι εδώ μιλάμε για δημόσια χρηματοδότηση. Πρέπει λοιπόν να δούμε επιπλέον ότι υπάρχει μια χρηματοδότηση η οποία έχει αποδοθεί σε ένα συγκεκριμένο ο κράτος μέλος και να ρωτήσω αυτό οφείλεται στο ότι ε, άλλα κράτη ακόμη δεν έχουν υποβάλει αιτήσει ή πρόκειται να υποβάλουν ή θα ανοίξετε αυτές τις δυνατότητες και σε άλλα κράτη-μέλη είναι ανοιχτή η δυνατότητα αυτή σε όλους. Ξεκινήσαμε το 2007 ε, με πολύ μικρή πρόοδο τα πρώτα χρόνια ε, γιατί εδώ μιλάμε για ε, νέα κράτη-μέλη. Βεβαίως ευχαρίστως να είχαμε και τα 27. Ε, και ήδη έχουμε πρώτες καλές ενδείξεις. Δεν θα έλεγα λοιπόν ότι ε, είναι αρνητική η εξέλιξη. Η Γερμανία συμμετέχει αλλά δεν μπορούμε τώρα να υπησέλθουμε σε λεπτομέρειες λόγω χρόνου. Ευχαρίστως να συζητήσουμε εκτός συνεδριάσεως. Η Γαλλία έχει επίσης ένα παρεμφερές μέσο, κάπως διαφορετικό και γι' αυτό βλέπετε λιγότερη συμμετοχή της Γαλλίας. Όσον αφορά τα δημοσιονομικά μέσα, ουσιαστικά αυτό το οποίο κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ό,τι προέρχεται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό είναι μία εγγύηση που παραμένει ως εγγύηση και ε, το μόνο που βλέπουμε είναι η αποτυχία, η αύξηση των επιτοκίων, πρόκειται δηλαδή ουσιαστικά ε, για χρήμα χρήματα τα οποία αντλούνται στην, ε, ε, ε, στη χρηματαγορά είναι όντως χρήματα τα οποία δεν είναι αποθέματα κάπου ή δημόσια χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Έλερ έχει ακόμη ένα διαδικαστικό. Ένα τεχνικό ερώτημα προς την Προεδρία. Τότε στον τριμερή διάλογο είχαμε συντάξει μία επιστολή η οποία παρουσίασε την δεύτερη δόση του προπολογισμού. Βέβαια τεχνικά αυτό είναι θέμα της Επιτροπής Προπολογισμού. Εμείς όμως ας ασχοληθήκαμε με αυτό τον τίτλο του προπολογισμού διακομματικά ο κύριος ε, Μπούζεκ τσίτσεστε και εγώ. Και το θέμα τώρα είναι πως ε, δεν δώσαμε λευκή επιταγή δηλαδή να υπάρξει μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση και μετά να δοθούν τα λεφτά αυτομάτως. Όχι, θα υπάρξει μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση και μετά θα αποφασίσουμε αν θα δοθούν τα χρήματα. Οπότε το ζήτημα τώρα τεχνικά είναι τι κάνουμε με αυτό το αντικείμενο εδώ πέρα. Μάλιστα, δεκτή η παρατήρηση. Θα το δούμε με τους συντονιστές στην επόμενη συνεδρία. Σας ευχαριστώ για την υπενθύμηση. Πιθανώς να μπει στην ε, επόμενη ημερήσια διάταξη. Θα το δει η γραμματεία. Είτε θα το συζητήσουμε με τους συντονιστές ή αν ε, ε θα μπει στην επόμενη ημερήσια διάταξη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Ερικα Μαν, τον κύριο Ζούτε. Καλή επιτυχία ευχόμαστε κτλ. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξη. Σχέδιο δράση για την ενεργειακή απόδοση και την αναθεώρησή του. Το έχουμε συζητήσει κάποιε φορέ. Τώρα έχουμε τις τροπολογίες και πολλή δουλειά βεβαίω για τον εισηγητή. Πολλές τροπολογίες σημαίνει μεγάλο ενδιαφέρον, κατοπιν καλό, αλλά σημαίνει και πολλή δουλειά. Κύριε Μπέντσεν, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση, είναι ένας αρκετά φτηνός τρόπος Η έκθεση ήδη συζητήθηκε από την Επιτροπή μας και έχουμε δει διεξοδικά αυτό το θέμα της ενεργειακής απόδοσης. Οι τροπολογίες είναι 428. Η έκθεση αυτή αφορά μία σειρά θεμάτων και γι' αυτό ε, ίσως ε, λόγω της εμβέλειας δηλαδή του θέματος έχουν ανακύψει τόσες τροπολογίες αυτό μας ενδιαφέρει είναι τα προϊόντα ενέργειας, οι πράσινες τράπεζες, τα μέσα μεταφοράς και ούτω καθεξής. Και υπάρχουν το, τροπολογίες που αφορούν το unbundling ως προς τους διάφορους παρόχους και νομίζω ότι αυτό το θέμα θα μπορούσε να δημιουργήσει αμφιγνωμίες ακόμα και για χώρες που θεωρούν ότι προηγούνται στον τομέα της απελευθέρωσης. Με τους σκιώδεις είδαμε ότι υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις σε σχέση με τους ε, στόχους της ενεργειακής απόδοσης. Υπάρχουν 17 τροπολογίες μόνο για την παράγραφο υπαριθμών 1, 7 τροπολογίες για έναν άλλο στόχο και γι' αυτό θεωρώ ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να φτάσουμε σε συμφωνία. Τα δεσμευτικά τμήματα της έκθεσης είναι πολύ σημαντικά θα πρέπει να υπάρχουν εγγυήσει από τα, ε, με βάση τους βασικούς στόχους. Το ΕΛΚ θεωρεί ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε αυτούς τους στόχους είτε είναι δεσμευτικοί είτε όχι. Και μετά από μία αποτίμηση από πλευράς κομισιών θα μπορούσαμε να προβάλλουμε μεμονωμένους στόχους για τα διάφορα κράτη-μέλη με βάση τα εθνικά σχέδια ενεργειακής απόδοσης. Επίσης υπάρχουν και οι προδιαγραφές. ένα ζήτημα το οποίο μας απασχόλησε. Μπορώ να σας πω ότι για την παράγραφο της παράγραφους 3 και 4 προσπαθούμε να συντάξουμε τροπολογίες συμβιβασμού. Στην παράγραφο 12 που αφορά τα κτίρια και εδώ υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις. Εγώ έχω προτείνει να επικεντρωθούμε στα δημόσια κτίρια των κρατών μελών, σχολεία και ούτω καθεξής. Οι φιλελεύθεροι και οι πράσινοι ζητούν να δούμε τα κτίρια στο σύνολό τους. Η παράγραφος αφορά την οδηγία για τις οικοπροβολές. Έχει μεγάλη σημασία να βελτιώσουμε την ε, ενεργειακή απόδοση. Έγινε λόγος λοιπόν για ενεργειακή σήμανση. Και πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε βασικές οικονομίες εάν έχουμε ε, οικοπροβολές, προβολές οικολογικού χαρακτήρα. Omkring finansieringsdelen ser det ud til, at der er største enighed i Ως προς την παράγραφο 24 μέχρι το τέλος του 2011 θα πρέπει να δοθούν ε, κίνητρα και νομίζω ότι μπορούμε να προωθήσουμε θέματα όπως ευφυείς μετρητές. Υπάρχουν ε, πρότυπα τα οποία μας ε, δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε, να προβούμε σε χρηματοδοτήσεις για να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Οι φιλελεύθεροι και οι πράσινοι ε, προέβαλαν τροπολογίες για τις πράσινες τράπεζες δεν έχω ολοκληρώσει το γύρο με τους σκιώδεις για αυτό το θέμα. Ε, βεβαίως θα πρέπει να βασιστούμε σε εμπειρογνώμενες που γνωρίζουν για τις πράσινες επενδύσεις αλλά και για τον τρόπο λειτουργίας του τραπεζικού τομέα. Εγώ προσπαθώ να φτάσουμε σε μία συνένεση. Θα πρέπει όμως να αποστείλουμε σημαντικά μηνύματα, διότι η ενεργειακή απόδοση μπορεί να βελτιώσει τις βιομηχανίες και την ανταγωνιστικότητα, ιδιαίτερα της ΜΜΕ, προβάλλοντας την ε, απασχόληση. Επειδή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τιμή ε, της ενέργειας τα επόμενα χρόνια. Μιλώντας για ενεργειακή πολιτική θα πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, ε, μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ πολιτικών ομάδων. Θα ήθελα να συνεργαστούμε για να φτάσουμε σε ένα συμβιβασμό έτσι ώστε να αποστείλουμε τα σωστά μηνύματα. So, jetzt habe ich eine Reihe von λοιπόν, τώρα έχει ζητήσει μια σειρά σαν Ξεκινάμε με του δύο ηγητές. Κυρία Τόμσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στις 12 Δεκεμβρίου 2008 και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ψήφισαν μια κρίσιμη απόφαση, την οδηγία περί ανανεωσίμων. Αποφασίσαμε πως το 2020 20% της κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Και βεβαίως η ανησυχία για η βάση αυτής της απόφασης ήταν η ασφάλεια της ε, παροχής ενέργειας. Και βέβαια ήταν ε, η αρχή μιας κοινή ενεργειακής πολιτικής και κυρίως οι μεγαλύτερες και ακριβότερες επενδύσεις στην ε, ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το οποίο αποφασίσαμε. Οπότε, το 20% δεν είναι ένα συγκεκριμένο νούμερο, είναι 20% ενός άλλου αριθμού που μεταβάλλεται. Οπότε έχουμε μια ευθύνη για την κατανάλωση ενέργειας. Για δεν πρέπει να αυξήσουμε τη σπατάλη της ενέργειας. Πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι, χρειαζόμαστε αποτελεσματική χρήση της ενέργειας για να γίνει η οδηγία των ανανεώσιμων όσο δυνατόν πιο φτηνή για τους πολίτες και να εξοδεύουμε λιγότερη ενέργεια. Για μένα είναι λογικό. Οπότε σαφώς η οδηγία αυτή των ανανεώσιμων πρέπει να ακολουθεί από μια ενέργεια για την ενεργειακή απόδοση και δεν αντιλαμβάνομαι γιατί είναι επίμαχο το αν θέλουμε να ξοδεύουμε λιγότερα για την ενέργεια και τις, την ασφάλεια προμήθειας ενέργειας. Γιατί είμαστε κατά των δεσμευτικών στόχων ενώ έχουμε δεσμευτικούς στόχους στην οδηγία για τις ανανεώσιμες Είμαστε πεπειραμένοι άνθρωποι εδώ πέρα, είδαμε τι έγινε στην οδηγία εδώ μέσα, τι συμβαίνει γενικά στις οδηγίες όταν δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Ήδη έχουμε μια οδηγία για 12% ενεργειακή απόδοση χωρίς δεσμευτικό στόχο. Και τι έχει γίνει, αυτό που έχει γίνει σε πολλές περιπτώσεις δεν πετύχαμε το στόχο. Εγώ ξέρετε πως είμαι Δανέζα δεν είναι πλέον έκτημα αυτό από μόνο του, αλλά στη Δανία από το 1979 δεν έχουμε ξοδέψει μία σταγόνα παραπάνω ενέργειας. Η κατανάλωση δηλαδή έχει μείνει η ίδια εδώ και 30 χρόνια. Γιατί οποιαδήποτε κυβέρνηση αριστερή, δεξιά, κεντρώα έχει ως στόχο την ενεργειακή απόδοση. Η οικονομία ανθεί. Δημιουργήσαν πολλές θέσεις εργασίας στον τομέα αυτών αλλά δεν σπαταλήσαμε περισσότερη ενέργεια. Και νομίζω πως μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτές τις ευκαιρίες της εμπειρίας μας στην Ευρώπη για να εξοικονομήσουμε και τα χρήματα των ανθρώπων. Νομίζω πως η ενεργειακή απόδοση είναι ένας τρόπος να πολεμήσουμε την ενεργειακή ένδυα. Άκουσα έναν βουλευτή της Ουγγαρίας που είπε πως τα νέα κράτη-μέλη 10% του πληθυσμού ξοδεύει 50% του εισοδήματός του το χειμώνα για να ζεστάνε τα σπίτια του. Ας κάνουμε λοιπόν τους στόχους ενεργειακής απόδοσης δεσμευτικούς, γιατί αλλιώς τα πράγματα δεν είναι λογικά. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπέντσιν για την εξαιρετική εργασία ε, ήταν τεράστια εργασία με τις 428 τροπολογίες και ε, είχε μία ιδιαίτερα συνεργατική προσέγγιση. Αύριο το πρωί και σήμερα θα συναντηθούμε εμείς οι σκιώδεις και νομίζω ότι πολλά μπορούμε να κάνουμε Uh, Νομίζω ότι θα πρέπει να φτάσουμε ε, σε συμπεράσματα και κατά την ελεύθερη μας εβδομάδα. Ίσως θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να φτάσουμε σε δεσμευτικούς στόχους, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι Υπάρχουν ε, άλλα ζητήματα. Και αυτό που έχει σημασία είναι να φτάσουμε σε ένα ουσιώδες αποτέλεσμα έτσι ώστε ο δημόσιος τομέας να δημιουργήσει μια πραγματική αγορά έτσι ώστε οι μικρές επιχειρήσεις να μπορέσουν να προωθήσουν υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης και ο ιδιωτικός τομέας θα αναλάβει αυτό το έργο όταν θα το έχει ολοκληρώσει ο δημόσιος. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα υπάρχοντα κτίρια, γιατί διαφορετικά το 2050 θα έχουμε κτίρια τα οποία θα δαπανούν τόση ενέργεια όση και σήμερα. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε την ανακαίνιση των ε, ήδη των κτηρίων. Συμφωνώ με τον ε, κύριο Πέντσεν σε σχέση με τους ε, μηχανισμούς αυτούς. Υπάρχει μία ανολοκλήρωτη εργασία της οδηγίας ε, που αφορά τα κτίρια και τη μόνωσή τους, νομίζω ότι θα πρέπει να προβούμε σε μια χρηματοδότηση, σε ένα σχέδιο χρηματοδότησης ενεργειακής απόδοσης, έτσι ώστε ε, οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν στις μεταφορές έχουμε ένα μεγάλο όγκο εργασίας. Ελπίζω να φτάσουμε σε λεπτομερείς ε, τροπολογίες συμβιβασμού και να έχουμε ένα λεπτομερές κείμενο με ρητές υποδείξεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να γνωρίζουν ποιες είναι οι προσδοκίες μας. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβάλλει συγκεκριμένες ιδέες πριν συνεδριάσουν στις 4 Φεβρουαρίου αρχηγοί κρατών. Και θα δούμε τι θα ανακύψει και από αυτή τη συνάντηση. Ο κύριος Ζαντώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να, να τονίσω την ποιότητα της συνεργασίας με κύριο Μπέντσεν και ελπίζω ότι θα είναι σαφές και στην τελική έκθεση αλλά αυτά που ακούμε τις τελευταίες εβδομάδες είναι πολύ θετικά. Νομίζω ότι ε, όπως πολύ σωστά είπαν οι συνάδελφοι σοσιαλιστές και φιλελεύθεροι ε, υπάρχουν ορισμένες ε, διαφορές απόψεων όσον αφορά τον δεσμευτικό χαρακτήρα της ενεργειακής κατάστασης. Ο κύριος Μπέντσεν ε, τόνισε τη θέση του ΕΛΚ. Τώρα σαν εισηγητής θα πρέπει να ε, εξεύρει μία συμβιβαστική λύση αποδεκτή για όλο το Κοινοβούλιο. Διότι πρόκειται εδώ για μία έκθεση κατά πρωτοβουλία η οποία καταρχήν πρέπει να στείλει ένα πολιτικό μήνυμα. Ξέρουμε ότι τη 4 Φεβρουαρίου θα έχουμε μια σημαντική διάσκεψη κολυφής στο θέμα αυτό και θα πρέπει να τεθεί ένα χρονοδιάγραμμα και αυτό προτείνουμε με τις τροπολογίες στον κύριο Μπέντσε να έχει ε, περισσότερο ένα χρονοδιάγραμμα και προθεσμίες για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα κατά τρόπον ώστε ε, η, να μπορέσει μπορέσει να υπάρξει και μία αναθεώρηση της ε, οδηγίας ε, για τις ενεργειακές υπηρεσίες πριν από το καλοκαίρι 2011 και θα πρέπει ε, εφόσον είναι μια έκθεση του Κοινοβουλίου να δίνει και ένα πολιτικό μήνυμα και σήμα και όπως συμφωνήσαμε τον κύριο Μπέντσεν ίσως η έκθεση αυτή δεν είναι πολύ φιλόδοξη. Το μήνυμα που δίνει για το 2020 δεν αρκεί. Θα πρέπει να συνδυάσουμε τις προτάσεις με ε, σαφείς στόχους για το 2020 αλλά και για το 2040 ελπίζοντας ότι ως τότε θα έχουν ανακαινιστεί όλα τα κτίρια πράγμα το οποίο θα αποτελέσει ένα ηχηρό μήνυμα που θα προέρθει από αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η κυρία Κολάνσκα Ροβίνσκα. Ευχαριστώ πολύ. Η εκθεσή μας είναι οπωσδήποτε ένα μήνυμα το οποίο μπορούμε να στείλουμε αλλά δεν θα ανακαινήσει τα σπίτια μία έκθεση. Αυτό τη φιλοδοξία των ε, στόχων μας. Ταυτόχρονα αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα. Το ότι δηλαδή δεν επιτυγχάνουμε τις υπάρχουσες ε, δεσμεύσεις. Σήμερα το πρωί μιλούσαμε για δεσμευτικούς στόχους και πρέπει να επιμείνουμε στόχους που έχουμε. Ο κίνδυνος είναι πως θα έχουμε τη μία έκθεση μετά την άλλη. Εγώ θεωρώ πως η Επιτροπή μας πρέπει να έχει μία άποψη, να μιλάει με μία φωνή, γιατί θα φαίνεται περίεργο το να λέμε το α στη μία έκθεση και το β στην άλλη. Με πολύ λεπτομερείς δεσμευτικούς στόχους. Οπότε εγώ θα επέμεινα και προτείνω να προσπαθήσουμε να είμαστε συνεκτικοί στη δράση μας. Δεδομένου του ότι ούτως ή άλλως θα συζητηθούν και οι δύο αυτές εκθέσεις τον Φεβρουάριο από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Όταν ε, μιλάμε για δεσμευτικούς ε, στόχους, Είχαμε πει ούτω ή άλλω πως θα είναι κάτι το δύσκολο να επιτευχθεί. Είναι φιλόδοξο στόχος, αλλά δύσκολο ε, να εφαρμοστεί. Γιατί δεν υπάρχει κοινή μεθοδολογία μέτρησης ενεργειακής αποτελεσματικότητας. Οπότε πώ θα μετρήσουμε το εάν έχει επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Θα πρέπει να θέτουμε δεσμευτικούς στόχους μόνο εάν είναι μετρήσιμοι. Δεν χρειαζόμαστε και άλλα κενά λόγια. Κύριος Σιμάνσκι. Ε, Ευχαριστώ. Η πολιτική μας ομάδα εκτιμά όχι μόνο την ε, μέθοδο συνεργασίας που επέλεξε ο εισηγητής, αλλά και με τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας. Όταν, δούμε, όταν βλέπουμε τις τροπολογίες συμβιβασμού, βλέπω ότι σε σχέση με τα, με τα στοιχεία, την, την ουσία των στοιχείων ε, αμφιγνωμίας, μπορούμε να ε, συγκλίνουμε ως προς την άποψη του εισηγητή. Νομίζω ότι θα πρέπει να κινηθούμε στα επιμέρους σε ιδιαίτερα ζητήματα. και δεν ορίζει νοερούς στόχους, δηλαδή καθαρά νοητικούς στόχους οι οποίοι δεν έχουν ένα έμπρακτο αντίκρισμα. Υπάρχουν όμως και πιο σοβαρά ζητήματα. Αν χρησιμοποιήσουμε την ε, ίδια μεθοδολογία, αν χρησιμοποιήσουν όλα τα κράτη-μέλη την ίδια μεθοδολογία, θα δουν ότι το κόστος της ενεργειακής απόδοσης θα επιμεριστεί διαφορετικά από τα διάφορα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν ε, ξεχωριστές καταστάσεις. Άρα ο συνδυασμός 7 που λαμβάνει υπόψη το σημείο εκκίνησης, δηλαδή την κατάσταση του κάθε κράτους μέλους, αποτελεί μια σημαντική προαπέτηση σε οποιοδήποτε κείμενο, διότι θέλουμε λύσεις που να είναι πραγματικά ε, δίκαιες, να έχουμε δηλαδή μια δίκαιη κατανομή του κόστους. Ιδιαίτερα σε κάτι τόσο σημαντικό όσο η ενεργειακή απόδοση. Η πολιτική μου ομάδα εκτιμά και τους, όλους, και τους άλλους τομείς ε, συμβιβασμού. Τη στιγμή που υπάρχει μία ε, σχετικά συσταλτική προσέγγιση ως προς την ανακαίνιση των κτηρίων, σε δείκτες της τροπολογίας 14, όλα αυτά μας ε, οδηγούν στο να έχουμε μια θετική εκτίμηση των τροπολογιών συμβασμού. Ευχαριστώ κύριε Σκυλακάκη. Mr. President. I would like to... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να στηρίξω τον συγκεκριτή στο θέμα των δεσμευτικών στόχων. Είναι σημαντικό αυτό. Γιατί αυτό το οποίο δεν λέμε συχνά είναι πως η ενεργειακή απόδοση δεν αφορά μόνο το θέμα της κλιματικής αλλαγής, ε, της ασφάλειας, ε, της ενεργειακής ασφάλειας, αλλά έχουμε και μία αποτυχία της αγοράς. Η ενεργειακή απόδοση, όσο έχει σήμερα σε κτίρια ή σε εταιρείε, δεν συμφέρει οικονομικά. Υπάρχει λόγος να παρέμβουμε, ακόμα και αν δεν υπήρχαν όλα τα ζητήματα που ανέφερα, η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή ασφάλεια. Επιπλέον, έχουμε και δουλειές που πρέπει να υπερασπιστούμε στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης. Όταν έχουμε δεσμευτικούς στόχους για τα ηλιακά πάνελ ή τις μιλάμε για βιομηχανικά προϊόντα, τα οποία πιθανότατα μετά από 10 χρόνια θα παραγόνται στην Κίνα. Και οι δουλειέ θα είναι στην Κίνα. Ενώ εάν βάλουμε δεσμευτικού στόχου για την ενεργειακή απόδοση, μιλάμε για δουλειέ οι οποίες θα μείνουν εδώ πέρα στην Ευρώπη. Οπότε υπάρχουν πολλοί λόγοι, οικονομικοί, περιβαλλοντικοί και λόγοι ασφάλειας ενεργειακής για να έχουμε δεσμευτικούς στόχους. Έχουμε δεσμευτικούς στόχους λοιπόν για τις ανανεώσιμες και όχι για την ενεργειακή απόδοση. Και δεν είναι λογικό αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως και όλοι εσείς διάβασα ε, προσεκτικά με συγχωρείτε τις τροπολογίες συμβασμού που πρότεινε ο κύριος Πένσεν, ο εισηγητής μας και θα ήθελα καταρχήν να τον ευχαριστήσω καθώς και τους σκιώδεις για την αφοσίωση με την οποία εργάστηκαν κατά τις ε, τελευταίες εβδομάδες. Άκουσα. Δύο λέξεις κλειδιά σήμερα το απόγευμα. Η Μπρίτα Τόμσεν μίλησε για λογική. Η δεύτερη λέξη ήταν η φιλοδοξία, ήταν η λέξη φιλοδοξία. Και είναι υπέρ και της λογικής και της φιλοδοξίας, αλλά υπό την ευρωπαϊκή έννοια, διότι η φιλοδοξία για μας ως ευρωβλεπτές σημαίνει ότι θα πρέπει αυτή η φιλοδοξία να συμμορφώνεται προς τις επιταγές της πραγματικότητας και λογική έχει, είναι πτυχή. Υπάρχει η χρηματοοικονομική σταθερότητα, η προστασία του περιβάλλοντος, η τεχνολογία, η πρόοδος τεχνολογίας. Υπάρχουν διάφορες οπτικές γωνίες της λογικής και μπρίτα. Δεν διαθέτει στο μονοπόλιο της λογικής νομίζω. Ας είμαστε φιλόδοξοι αλλά κατά τρόπο ώστε να συμμορφωνόμαστε προς τις επιταγές πραγματικότητες. Και η, λογική είναι ε, πολύ σήμαντη και κανένας διαθέτει το μονοπόλιο της ε, λογικής. Καλωσορίζω τις τροπολογίες συμβιβασμού, το συμβασμό που προβάλλεται στις τροπολογίες σε σχέση με την πρόθεση του CHP. Καλύτερη αποδοτικότητα ως προς την θέρμανση και για την ομάδα μου ύψης της σημασίας είναι το CHP. Αυτό αφορά και την ε, κτηρίων και ούτω καθεξής. Και για την παράγραφο 1 δέχομαι την τροπολογία συμβασμού, διότι η πρόταση αυτή είναι πραγματικά φιλόδοξη και προβάλλει μία εις βάθος αξιολόγηση της κατάστασης και αυτό σημαίνει βραχυχρόνιες προσπάθειες έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε βήματα προς τα εμπρός για την ενεργειακή αποδοτικότητα ενώ του Συμβουλίου Ενέργειας της 4 η Φεβρουαρίου. Και επειδή η παράγραφος αυτή έχει διατυπωθεί κατά τρόπον ώστε να αφήνει περιθώρια ελιγμού για τον καθέναν αφού η Επιτροπή θα έχει δημοσιεύσει αυτή την αξιολόγηση. Πιστεύω ότι το πρόγραμμα δράσης μας δίνει τις κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές για να ξέρουμε πώς και πότε θα να φτάσουμε σε αυτούς τους στόχους για την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά 20% μέχρι το 2020. Ως προς τους μεμονωμένους στόχους έχουμε την κατάλληλη ευελιξία. Μπορεί κανείς να δράσει ως προς τη διαδικασία. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων. Και υπάρχει ένα σημείο στο οποίο θα ήθελα να επιμείνω. Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης για να φτάσουμε στους στόχους ε, αποδοτικότητας, αυτό αποτελεί κάτι το επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνη προσέγγιση. Όταν μιλάμε για απόδοση, μιλάμε περισσότερο output με λιγότερο input. Να είμαστε πολύ σαφείς ως προς αυτό ως προς αυτή την ενιολογική βάση. Αν θέλουμε μία ανταγωνιστική ε, αγορά, η απόδοση είναι σημαντική, αλλά η μείωση κατανάλωση σε απόλυτους όρους ίσως έρχεται σε αντίφαση με αυτό. Δεν θα πρέπει να δεχόμαστε ιδεολογικές ε, ιδεολειψίες. Είμαστε Ευρωπαίοι Ευρώπη σημαίνει συνένεση, σημαίνει ε, ε, συμφιλίωση ε, αποκλίνουσων απόψεων και αυτό αποτελεί και αυτή την πρόταση. Είναι μια πρόταση συνένεσης. Είναι δε τόσο λογική που σήμερα το πρωί την δεχτήκαμε στην έκθεση Μπομπίνσκα Άρα θα έρθουμε σε αντίφαση με, σε μια έκθεση που ε, εκπληρώνει ένα σκέλος της γενικής εμβέλειας έκθεσης. Κανένα δεν θα μας πάρει στα σοβαρά. Σήμερα το πρωί εγκρίναμε μια πρόταση και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να είμαστε συνεπείς με αυτό που εγκρίναμε σήμερα το πρωί. Ευχαριστώ και δίνω το λόγο στον κύριο Πίπερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Την τελευταία εβδομάδα είχαμε αποφασίσει στο, την περασμένη εβδομάδα αποφασίσαμε στο Κοινοβούριο ότι θα ενθαρρύνουμε ε, τους ε, καταναλωτές ε, ε, ε, τους επιχειρηματίες να πληρώνουν τους μισθούς, τους κατώτατους μισθούς και τώρα ζητούμε να περικόψουμε την ενεργειακή κατανάλωση. Πώς θα δημιουργήσουμε όμως θέσεις εργασίας. Αυτό μας ενδιαφέρει για να μην έχουμε έχουμε ε, άλλα προβλήματα αλλά δεν, θέλ, δεν αστείευομαι τώρα νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα όριο και με αυτά τα ποσοστά απλούστατα μας ξεφεύγουν τα έξοδα και το βλέπουμε και στα κράτη-μέλη και εις τις επιχειρήσεις που οπλίτονται και στις οικογένειες που χρειάζεται να πληρώσουν πιο ακριβά την ενέργειά τους και πρέπει να βρεθεί ε, μία στρατηγική που να δεσμεύεται να μειώσει το κόστος της ενεργείας και όπως ελέγχθη πολύ σωστά έχουμε μεν μία στρατηγική η οποία έχει συζητηθεί μέχρι το 2020 που έχει πολύ έξυπνες πτυχές και μας έχει σχεδιαγραφίσει πολλές δυνατότητες και τέλος εγώ θα ήθελα να πω ότι μπορούμε να κάνουμε ε, με αυτούς τους στόχους διότι υπάρχει κάτι έξυπνο σε αυτά που είπε ο κύριος Μπέντσεν ε, δεν έχει αξιολογηθεί ε, εάν τα δεδομένα τα οποία δημιουργήσαμε έχουν εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο διότι υπάρχουν ατελείωτες ευρωπαϊκές δυνατότητες να ε, ελέγξουμε περισσότερο την ε, κατάσταση προτού θέσουμε άλλους δεσμευτικούς στόχους. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε που αναφέρονται εις ε, την έκθεση αυτή και γι' αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να οξύνουμε την νομοθετική μας εργασία αλλά να είμαστε πιο δημιουργικοί. Ο κύριος Γκέρεκ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, σύντομα θα ήθελα να πω και εγώ δύο λόγια για την ε, έκθεση Μπέντσεν. Συμφωνώ με την διαφοροποιημένη προσήγηση σε διάφορες ε, χώρες γιατί κάθε χώρα χρειάζεται μια διαφορετική λύση γιατί υπάρχει διαφορετικό πεδίο οικονομικής ανάπτυξης. Όμως όσον αφορά τα κτίρια Ίσως οι δυτικοί συνάδελφοι δεν ξέρουν πάρα πολλά γι' αυτό, αλλά στα νέα κράτη-μέλη και στη χώρα μου, στην Πολωνία, στη Ρουμανία, τη Σλοβακία, την Τσεχία, έχουμε πολύ μεγάλες πολυκατοικίες, ε, εργατικές κατοικίες που θα μπορούσαν να εξυγχρονιστούν για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση. Αυτό ίσως ε, δεν έχει γίνει ε, αντιληπτό από αυτά τα οποία λέει ο εισηγητής. Ο καλύτερος τρόπος βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης είναι μέσω της τεχνολογίας. Υπάρχει μια οικονομική και μια τεχνολογική πτυχή. Θεωρώ λοιπόν πως οι περισσότεροι εστιάζουν πάρα πολύ στην, ε, στην οικονομική πτυχή. Η τεχνολογική όμως απόδοση είναι κλειδί εδώ πέρα, δηλαδή πόσο ποστό της ενέργειας καταλήγει όντως σε παραγόμενο έργο. Δυστυχώς όμως πρέπει να πω πως το πακέτο ενέργειας και κλίματος που υιοθετήσαμε πέρσι και ειδικά η έκθεση Davis για την δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξη ενέργειας από άνθρακα, κάτι το οποίο δεν αντιλαμβάνομαι γιατί ο άνθρακας είναι εξαιρετικά αποδοτικός. Μιλάμε για ένα 60 μέχρι και 70, ίσως και 80% ενεργειακή απόδοση. Οπότε σας παρακαλώ να το ξαναδείτε αυτό, γιατί αυτό το οποίο ζητάμε είναι να συμβουλεύσουμε την Κομισιόν. Εγώ λοιπόν προτείνω να το κοιτάξουμε αυτό. Κύριε Τόμσεν, πράγματι υπάρχει ενεργειακή φτώχεια, αυτό είναι αλήθεια και στη χώρα μου 40% των δαπανών των οικοκυριών πηγαίνει στην ενέργεια. Δεν είναι 10% όπως στη Δυτική Ευρώπη, 40% Σκεφτείτε το και αυτό. Σας ευχαριστώ κύριε Φανίστελ Ροδί. Σας ευχαριστώ και εγώ ε, σας ευχαριστώ για αυτή την ε, έκθεση είχα την αίσθηση πως ε, πάμε σε μια νέα φάση, πως φεύγουμε από τους δεσμευτικούς ε, στόχους και μπορούμε να δούμε τα διάφορα μέσα ε, έτσι ώστε τα, τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να, να συνεισφέρουν και να κρίνουν εκείνα ποια είναι τα μέτρα με τα οποία θα μπορέσουν να εκπληρώσουν τα διάφορα κριτήρια και να καταρτήσουν τα κράτη-μέλη τα, σχέδια αυτά. Και εντάξει, γεγονό είναι πω τα κριτήρια θα πρέπει να τεθούν αυστηρότερα στη διαπραγμάτευση μεταξύ Κομισιών και κρατών μελών. Και να υπάρχουν μετά μεμονωμένοι στόχοι. Και νομίζω πως ε, η λογική του κυρίου Βιδάλ Κουάδρας νομίζω είναι η ε, σωστότερο. Εγώ θέλω λοιπόν να σκεφτούμε περισσότερο για το πώς θα μπορέσουμε να δούμε και να υπολογίσουμε τα εθνικά σχέδια ενεργειακής απόδοσης και εκεί πέρα νομίζω υπάρχει η ε, καινοτομία. Πρέπει να έχουμε νομίζω να δείξουμε και κάποια εμπιστοσύνη και η τεχνολογία μας εξυπηρετεί εδώ πέρα και μπορούμε πράγματι να επιτύχουμε πάρα πολλά πράγματα. Αυτό δεν γίνεται μόνο με κεντρικά δεσμευτικά ε, κριτήρια σας ευχαριστώ. Κύριε Μπέντσεν, θέλετε ξανά τον λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως ακούσαμε πολλά ζητήματα και θετικά σχόλια ακούστηκαν και στη συνέχεια θα εργαστούμε πολύ σκληρά. Πρέπει να διανύσουμε μεγάλο δρόμο πριν βρούμε ε, ένα ε, κοινό παρονομαστή για την Επιτροπή μας. Θα το προσπαθήσω αυτό. Έχει μεγάλη σημασία για την ανταγωνιστικότητα, για το μέλλον και για να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τα θέματα, θα προσπαθήσουμε να τα επιλύσουμε πριν από την, την επόμενη συνάντηση και τις επόμενες μέρες θα συναντηθούμε τους Κιώδης. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, λέει ο Πρόεδρος. Οπότε περνάμε στο επόμενο. Ναι, τις προθεσμίες τις ξέρετε. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα για τροπολογίες και 9 Νοεμβρίου η ψηφοφορία. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι κρατικέ ενισχύσει που διευκολύνουν την πάυση λειτουργία μη ανταγωνιστικών ανθρακοριχείων. Ο συνάδελφο Ζαντό είναι εδώ πέρα εισηγητή. Έχετε τον λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό. Ξέχασα να ρωτήσω για την ε, ενεργειακή αποτελεσματικότητα αν είχε να σχολιάσει κάτι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με συγχωρείτε κύριε Ζαντό, το ξέχασα, σας ζητώ συγγνώμη και δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα είμαι πολύ σύντομη. Καταρχήν, σας ευχαριστώ για το σχέδιο αυτό εκθέσεως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα το παρακολουθήσει με πολύ προσοχή είναι ενδιαφέρον διότι συνάδει με το σκεπτικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίσης καλό θα ήταν να σας αναφέρω ότι είναι πολύ επίκαιρο θέμα και έχει θαυμάσιες δυνατότητες να ε, προωθήσει τις ιδέες ε, της ΙΤΡ που θα ληφθούν υπόψη στον προγραμματισμό και την αποτελεσματικότητα που προβλέπονται. Θα το θα το επεξεργαστούμε με στόχο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Αρχών ε, ε, Φεβρουαρίου και ήδη θα έχετε ε, δει τις πρώτες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στρατηγική 2020 που αναφέρεται στην ενεργειακή αποτελεσματικότητα και όπου θα δούμε πώς η στρατηγική αυτή μπορεί να αναπτυχθεί με περισσότερες λεπτομέρειες. Σας ευχαριστώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσβλέπει στην ε, ε, ε, εξέταση της πλήρους εκθέσεως. Ευχαριστώ πολύ, με συγχωρείτε που τους ξέχασα. Κύριε Ζαντό, τώρα έχετε το λόγο. Και ε, χρησιμοποίησαμε το διάλειμμα για να γράψουμε πολλούς οι οποίοι ζητούν το λόγο. Να σας υπενθυμίσω λοιπόν ότι για το φάκελο αυτό είχαμε συζητήσει, συναντηθήκαμε τους σκιώδεις εισηγητές, αρκετά επικοδομητικές συζητήσεις και ανταλλάξαμε απόψεις και με μηνύματα ηλεκτρονικά και νομίζω ότι σε ορισμένα θέματα έχουμε προχωρήσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει μία πρόταση για τη ρύθμιση. Συζητάμε ε, τις ε, ε, κρατικές ενισχύσεις για την πάση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών επιχειρήσεων και στο Συμβούλιο θα χρειαστεί ομοφωνία για να τροποποιηθεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την πρώτη λανθασμένη αντίληψη που πρέπει να διευκρινίσουμε για να μην πάρει κακό δρόμο η συζήτηση είναι ότι δεν προτείνουμε εδώ να κλείσουμε με τα ανθρακορικεία ή τις, ε, και, ε, τις, ε, τους ηλεκτρικούς σταθμούς που χρησιμοποιούν άνθρακα και αφήνει ε, στα κράτη την ε, ε, ελευθερία επιλογής του μείγματο που θα χρησιμοποιήσουν για την ενέργεια. Απλώ αναφέρεται στο κλείσιμο των ανθρακορικίων που δεν είναι ανταγωνιστικά και στις προϋποθέσεις της, της επάυσεως λειτουργίας τους και αν αφαιρόμαστε ή στην Ισπανία που είχαν λάβει από το 1995 7 ε, ε, ε, αναβολές για την χρησιμοποίηση εθνικών ενισχύσεων που προβαίνουν σε το ανταγωνισμό στον άνθρακα της Πολωνίας και ε, ο οποίος είναι παραδείγματο χάρη 8 φορές λιγότερο δαπανηρός από ότι ε, το ισπανικό κάρβουνο. Άρα δεν κλείνουμε τα ανθρακορικεία ούτε τις, ε, τους σταθμούς οι οποίοι χρησιμοποιούν άνθρακα. Το δεύτερη λανθασμένη αντίληψη. Δεν αναφερόμαστε εδώ στις αποτελεσματικές τεχνολογίες που άπτονται του άνθρακα γίνονται συζητήσεις για καθαρό άνθρακα, αλλά δεν είναι το θέμα που μας απασχολεί σε αυτή τη ρύθμιση. Απλώς θέλουμε να παρακολουθήσουμε τις μη και τα μη ανταγωνιστικά άνθρακορίσικια. Υπάρχουν άλλες έρευνες σχετικά με τον άνθρακα και τον χάλευρα ή με το ETS που αναφέρονται στις τεχνολογίες που συνδέονται με τον άνθρακα και κάθε φορά προσπάθησα να χρησιμοποιήσω τροπολογίες επί των συζητήσεων που είχαμε για να διευκρινίσω τα σημεία αυτά. Αυτή η ρύθμιση θα μπορούσε να αναφέρεται σε επενδυτικές ενισχύσεις. Εδώ δεν θέλουμε να επιτρέψουμε στα κράτη να επενδύσουν στο άνθρακα αλλά απλώς επαναλαμβάνω να καλύψουμε την πάυση λειτουργία των μη ανταγωνιστικών ανθρακορικίων μέχρι το 2014 αν υπάρχουν ενισχύσεις ε, ε, για, ε, για το κλείσιμο και μέχρι το 2026 εάν υπάρχουν κοινωνικές πτυχές της πάυσεως λειτουργίας. Επίσης πρέπει να δούμε τι γίνεται με τον τομέα όταν υπάρχει μία πτώσεις και ε, ε, αυτό έχει γίνει και για την κλωστοϊφαντουργία. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε ε, κάθε δυνατότητα προσανατολισμού των εργαζομένων, ιδίως στις περιοχές όπου υπάρχουν μόνο βιομηχανίες και να δούμε τι άλλες βιομηχανικές εναλλακτικέ λύσεις υπάρχουν όταν ο άνθρακας δεν είναι ανταγωνιστικός και πώς θα εστιάσουμε τη συζήτηση συζήτηση για να αποφύγουμε το κλείσιμο αυτών των ορυχείων να οδηγήσουν σε ε, μία ερήμωση της περιοχής. Τώρα, αυτό το οποίο παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι, ε, ε, οι διάφοροι επίτροποι δηλαδή είναι μια συμβιβαστική λύση διότι οι πράσινοι συνάδελφοι θα ήθελαν να σταματήσει το καθεστώς αυτό από το 2010 να σταματήσουν άμεσα οι κρατικές ενισχύσεις και απλούστατα να ασχοληθούν με την αναδιάρθρωση και τον επαναπροσανατολισμό των εργαζομένων αλλά ξέρετε ότι υπάρχουν λεπτές ε, υπηρεσίες, λεπτές ισορροπίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο. Δεν συζητάμε πώς θα χρησιμοποιηθεί το κάρβουνο την επόμενη 20 ετία, αλλά πόσο θα καλύψουμε μη ανταγωνιστικά ανθρακοριχεία και ξέρετε ότι το 2014 είναι ε, μια συμβιβαστική λύση και όχι οικολογική ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ότι ο συμβιβασμός αυτός μπορεί να σημαίνει ακόμη και μεταξύ επιτρόπων ότι θα οδηγηθούμε σε ε, μία απουσία ρυθμίσεως μετά το 2010. Γι' αυτό, αυτό λέγουν οι τροπολογίες. Ζητάμε για τις ε, μονοβιομηχανίες προγράμματα αναπροσανατολισμού να υπάρξει η χρηματοδότηση στις ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας και να συνεχίσουμε να σεβόμαστε την αρχή ότι ο Ριπένον πληρώνει και όταν υπάρχει κρατική ενίσχυση δεν δίνουμε, δεν χρηματοδοτούμε τις επιχειρήσεις οι οποίες κερδίζουν και από αλλού. Οι κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να ασχοληθούν μόνο ε, με τους ε, μη ανταγωνιστικούς τομείς στη μεταβατική περίοδο και να μην αντικαταστήσουν τα κέρδη των ε, επιχειρήσεων σε άλλους τομείς. Ε, με συγχωρείτε, ε, αλλά ελπίζω ότι έπρεπε να επεκταθώ λίγο παραπάνω για να είναι σαφής η συζήτηση που θα έχουμε στη συζήτηση. Κυρία Ρέρα Μαντουρέλ καταρχήν. Ο κύριος Σέντσου θα ήταν καλύτερα να λάβει το λόγο πρώτα γιατί ε, μιλά εξ ονόματος της Σκιωδούς. Ο κύριος Σέντσου έχει το λόγο. Η κυρία Τσικάου είναι η Σκιώδης και ζητά συγγνώμη γιατί δεν βρίσκεται εδώ. Γι' αυτό μιλώ εξ ονόματός της. Ο άνθρακας έχει μεγάλη σημασία στον ενεργειακό τομέα. Χρησιμοποιείται κατά 30% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Γερμανία μόνο 7,2%, στη Γερμανία κατά 40%. Όμως τα άνθρακοχεία ε, διασφαλίσουν 238.000 θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα σε μονοβιομηχανικές ζώνες. Το, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε εισαγάγει εκατομμύρια ε, ε τόνους ε, άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για τον ευρωπαϊκό ισολογισμό, για το ισοζύγιο πληρωμών μας μάλλον. Γι' αυτό θα πρέπει να διασφαλίσουμε τις ε, μεγαλύτερες δυνατές ποσότητες. Χωρίς τις κρατικές ενισχύσεις θα μειωθεί η παραγωγή μας κατά 20% και θα μειωθούν οι θέσεις εργασίας κατά 100.000 οι κρατικές ενισχύσεις έχουν ε, μειωθεί από 6 δις σε 2,9 δις το 2009. Θεωρούμε ότι οι κρατικές ενισχύσεις είναι αναγκαίες για να παραμείνουν τα άνθρακα ανταγωνιστικά. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να είναι ανταγωνιστικά τη στιγμή που δεν διαθέτουν ε, τεχνολογίες εχμής. Θα πρέπει να εξυγχρονιστούν. Η διαδικασία εξυγχρονισμού και η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας είναι μια ε, μακροχρόνια διαδικασία. Δεν εξασφαλίζεται εν μία νυχτή για να υπάρχει σωστή εκμετάλλευση θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το άρθρο 3F και να μειώσουμε το ποσοστό κατά 10% και βεβαίως να κλείσουν τα ανθρακοριχεία που δεν είναι ανταγωνιστικά. Αλλά αντί για το 2015, στο 2022, διότι θεωρούμε ότι ε, έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Δεν θα πρέπει παρά να κλείσουν τα ανθρακοριχεία που δεν είναι ανταγωνιστικά. Θα πρέπει ο όμως να βοηθήσουμε τα ανθρακοριχεία να γίνουν ανταγωνιστικά εκεί που είναι δυνατόν. Θα ήθελα να μου διασαφηνίσει κάτι, Επιτροπή. Μιλάμε για τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, μπορεί να ε, μειωθεί αυτή η προθεσμία, δηλαδή να επαναπροσδιοριστεί. Ματουρέλ, θα ήθελα να πω ότι ε, θα πρέπει να πω ότι το κλείσιμο το μη ανταγωνιστικών ανθρακοριχείων θα πρέπει να γίνει μέχρι το 2020 ή 2022 διότι θα υπήρχαν πολύ αρνητικές οικονομικοκοινωνικές συνέπειες. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε πολλές περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα ανθρακοριχεία αποτελούν μεγάλη πηγή εισοδήματος. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει το θέμα του περιβάλλοντος και γι' αυτό η Επιτροπή πρότεινε ως προθεσμία το 2014. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανεργία, την απώλεια θέσεων εργασίας και την παρεπόμενη φτώχεια που θα δημιουργεί το εάν ίσχυε το 2014 για αυτές τις περιφέρειες που δεν έχουν το αναγκαίο χρονικό διάστημα για να προβούν σε αυτό τον ε, επαναπροσδιορισμό. Υπάρχουν και δύο άλλα σημεία. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει ένας επαναπροσδιορισμός αυτών των περιφερειών Γι' αυτό θα ήθελα οι ευρωπαϊκές αρχές να επαγρυπνήσουν έτσι ώστε ο εισαγόμενος άνθρακας να πληρεί τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους που προαπαιτούνται από τον ευρωπαϊκό άνθρακα. Αυτή θα είναι μία, μία από τις τροπολογίες μου και θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνουν και οι κατάλληλες επενδύσεις για την μείωση των ρήπων και γι' αυτό θα υποστηρίξω οποιαδήποτε τροπολογία υπό αυτή την έννοια. Ευχαριστώ. Κύριος ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Κάποια σχόλια και μια ερώτηση προς την Κομισιόν. Πρώτο σχόλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να εκμεταλλευτεί το ότι εκπνέει ο προσωρινός ε, κανονισμός. Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνο γι' αυτό. Προφανώς η Κομισιόν θέλει να σταματήσει τελείως η ε, εξόρυξη άνθρακα. Είναι δογματική και τρελή αυτή η προσέγγιση. Αυτό θα δημιουργήσει μοιραία σε αθέμητο ανταγωνισμό. Οπότε το ερώτημά μου είναι γιατί να μην, γιατί να μην αυξήσουμε τους δασμούς ε, σε εισαγωγές άνθρακα από τρίτες χώρες. Αυτή είναι υπεύθυνη για το ότι είναι μη ανταγωνιστικός ο δικός μας άνθρακας, ε, ο δικός τους επιδοτείται. Στην Πολωνία έχουμε έλλειψη επενδύσεων. Σήμερα πέθανε ένας ε, ανθρακορίχος στην Πολωνία. περνάμε σε μια κατάσταση στην οποία θα έχουμε έλλειψη ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη. Θέλω πραγματικά ποιος είναι ο στόχος της Κομισιόν να καταστρέψει τον άνθρακα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος συγητής εδώ πέρα μίλησε για κάποια λάθη στη βάση αυτής της συζήτησης. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω άλλο ένα λάθος. Γιατί η Κομισιόν αγνόησε τους εθνικούς συμβασμούς ε, αφαίρετα ενώ π.χ. στη Γερμανία έχουμε φτάσει στο 2018 ε, και η Κομισιόν κατέληξε το 2014. Το λόγος δεν είναι το δίκαιο του ανταγωνισμού, δεν είναι τόσο ελάχιστα τα ποσά που δεν μπορούμε να μιλάμε για στρέβλωση. Ο στόχος και το είπε η Κομισιόν ανοιχτά είναι πως για λόγους προστασίας του κλίματος πρέπει να τελειώσει αυτή η τεχνολογία του στομότερο δυνατόν. Και αναρωτιέμαι τι θα γίνει εάν στην όλη αυτή αλυσίδα παραγωγής ενέργειας, ορυχείο και παραγωγή ρεύματος βγάλουμε το ορυχείο από τη μέση. Τι θα γίνει, θα εισάγουμε το άνθρακα, τον άνθρακα από την Κίνα. Και αν λάβουμε εμεί την απόφαση να το κλείσουμε το 2014 και εξακολουθούν τα εργοστάσια παραγωγή ρεύματο να λειτουργούν άλλα 20 χρόνια, η μεταφορά του άνθρακα από πλευρά κλίματο είναι ούτω ή άλλω καταστροφική. Αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο λάθο στο οποίο εξαναγκαζόμαστε. Εξαναγκαζόμαστε να κάνουμε πράγματα τα οποία έχουν κάποια πιθανότητα ίσως να επικοινωνήσουν, να λειτουργήσουν τα ορυχεία αυτά. Οπότε έχουμε πέρα του 2018 και θα ζητήσω και το 2020 και θα ήθελα να πω και το εξής. Εγώ ζω σε 10 χιλιόμετρα από ένα ανθρακοριχείο το οποίο βρίσκεται ελάχιστα απέχει από το να είναι ανταγωνιστικό. Εάν πει ένας επενδυτής πως εγώ θέλω να επενδύσω εδώ πέρα επειδή θα ανέβουν οι τιμές της ενέργειας και αυτό είναι για μένα μια μεγάλη ευκαιρία για μένα, πρέπει τουλάχιστον να δώσουμε την δυνατότητα να υπάρξει μια χρηματοδότηση στον τομέα της ε, ενεργειακής απόδοσης και να επιτρέψουμε σε αυτούς τους ε, επενδυτές να κάνουν αυτή την πιθανή επενδύση. Οπότε αυτά τα δύο πράγματα, 2018-2020 και η δυνατότητα ιδιωτών επενδυτών να μπορέσουν να εμπλακούν. Αυτά και, ε, τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά για μένα. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Μακινιέβιτ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, το 2010 είναι το τελευταίο έτος του κανονισμού για τον άνθρακα σχετικά με την ανταγωνιστικότητα των ε, ορυχείων, όπως επίσης και την εγγύηση της ενεργειακής ε, ασφαλείας. Η αποδοτικότητα εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Μπορούμε δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε διάφορους ορισμούς. Εγώ προέρχομαι από μία περιοχή που βασίζεται εις τα ανθρακοριχεία και από εκεί παράγεται ένα μεγάλο μέρος ε, ο άνθρακα ο οποίος χρησιμοποιείται για ηλεκτρισμό. Άρα ο άνθρακας ε, αποτελεί ένα βασικό παράγοντα της ε, παροχής ενεργείας. Η ε, παραγωγή έχει διπλασιαστεί και η πρωτογενής παραγωγή θα διπλασιαστεί, δηλαδή θα είναι μεγαλύτερη από του πετρελαίου και ε, αν ε, χρειάζεται αυτός ο άνθρακας στην Ευρώπη ε, θα κλείσουν τα ανθρακοριχεία γιατί τότε σε 20 χρόνια θα πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει ότι οι ανάγκες θα παραμείνουν σταθερές. Θα χρειαστεί τότε να εισάγουμε γι' αυτό και πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει συγχρηματοδότηση των προσπαθειών των κρατών μελών για να χρησιμοποιηθούν νέες τεχνολογίες και να εξασφαλίσουμε μία ενεργειακή σταθερότητα στα κράτη και για να μπορούμε να επιτύχουμε τους φιλόδοξους στόχους της στρατηγικής του 2020. Όσον αφορά την ρύθμιση την οποία συζητάμε, μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν κράτη τα οποία βασίζονται στην χρήση του άνθρακα και το ρητό μάλλον η απόφαση του Συμβουλίου του 2007 επιτρέπει σε κάθε κράτος να αποφασίσει πόσο θα διαμορφώσει το ενεργειακό του μείγμα ε, και ε, γι' αυτό θα πρέπει τα ε, κράτη να μην οδηγηθούν εις τον αποκλεισμό του άνθρακα από το ενεργειακό μείγμα θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει μία σωστή αντιμετώπιση και εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε οι ενισχύσεις να μην καλύπτουν μόνο 20% αλλά 30% και όσον αφορά τις ενισχύσεις για την πάυση λειτουργίας ε, στην, ε, θα έπρεπε να σταματήσουν την 1η Οκτωβρίου 2020 θα ήθελα εδώ να αναφερθώ εις ε, τα σχόλια του εισηγητή, διότι αυτός ε, αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα ε, που συζητήθηκαν μεταξύ σκιωδών εισηγητών. Για μας το, ο άνθρακας είναι ε, συνδεδεμένος με την Τσεχία και με την πάυση λειτουργίας και γι' αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει ε, όλα τα ε, θέματα να ε, εξεταστούν σφαιρικά και γι' αυτό θέσαμε τόσα πολλά. Ο κύριος Χατζημαρχάκης. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τον εισηγητή για την πολύ σωστή και δικαιή πρόσκληση των σκιωδών εισηγητών και για το ότι μοιράστηκε τις γνώμες μας. Βεβαίω δεν τίθε ζήτημα πω τα μη ανταγωνιστικά ανθρακοριχεία πρέπει να κλείσουν. Αυτό είναι κάτι που θα γίνει μακροπρόθεσμα. Το θέμα είναι πότε λοιπόν θα τελειώσουν οι επιδοτήσει. Και το γεγονό πω ο επίτροπο Αλμούνια, ω ε, ανώτατο εκπρόσωπο του ανταγωνισμού στην αρχή του πρόταση, ε, πρότεινε το 2020 και το 2022 ακόμα, δείχνει πως, όπως είπε και ο κύριο Πίπερ, το μεγαλύτερο ζήτημα δεν είναι ο ανταγωνισμό, είναι ένα πολιτικό ζήτημα το οποίο το χειρίστηκε πολιτικά το σώμα των Επιτρόπων και ενάντια της άποψης μάλιστα του Προέδρου και του Επιτρόπου Ανταγωνισμού. Πάρα πολλά κράτη-μέλη μετά από αγώνα οδηγήθηκαν σε κάποιες συμφωνίες ε, το 2018 για την Γερμανία. Ως φιλελεύθερος εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος για το ότι θα ενισχύουμε επί τόσο καιρό, αλλά τώρα το έχουμε ορίσει ε, υπάρχουν πάρα πολλές συμβάσεις που βασίζονται σε αυτό και πάρα πολλές μεταβατικές διατάξεις και μάλιστα ένας τερματισμός της επιδότησης το 2014 θα μπορούσε και θα οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος από ότι να εξαντληθεί ε, η επιδότηση το 2018 και δεν μπορούμε να το πούμε αυτό στους φορολογούμενους. Πώς εξηγείται αυτό. Από τα λεγόμενα διαρκή κόστη, το κόστος ιονιότητας όπως λέγεται. Δηλαδή, εάν μεταβούμε σε άλλες ε, πηγές ενέργειας θα πρέπει να οδηγηθούμε σε νέες ε, συνδέσεις. Ε, δηλαδή, ένα ανθρακοριχείο το οποίο έχει κλείσει θα πρέπει να δημιουργηθεί, να οδηγηθεί σε μια κατάσταση και αυτό έχει πολύ συγκεκριμένες διατάξεις οι οποίες ε, εάν το πάμε ε, εις άτοπον οδηγούμαστε στο ότι το 2018 συμφέρει περισσότερο από το 2014 τελευταίων. Πριν από λίγες ημέρες πανηγυρίζαμε όλοι για την απελευθέρωση κάποιων ανθρακορίχων στη Χιλή που πέρασαν μήνες στο σκοτάδι και μπόρεσαν να δουν ξανά το φως σήμερα. Η τεχνολογία αυτή είναι γερμανική και δεν θα υπήρχε εάν δεν υπήρχαν ενισχύσεις στη Γερμανία. Υπάρχει λοιπόν εδώ πέρα μια πτυχή έρευνας και καινοτομία που πρέπει να δούμε. Είμαστε πρώτοι ε, πρώτες οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε πάρα πολλούς τομείς και αν τα διαγράψουμε όλα αυτά από τη μια μέρα στην όλη θα έχουμε χάσει αυτό ε, τον ηγετικό μας ε, ρόλο. Δεν μιλάμε δηλαδή μόνο για μια πεπαλαιωμένη και τελειωμένη τεχνολογία, αλλά και για τελείως καινοτόμες τεχνολογίες. Γι' αυτό θα υποστηρίξω και εγώ αυτήν την τροπολογία για το 2020. Σας ευχαριστώ. Να δώσω λόγο στον κύριο Ράμζοφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τρία σημεία θα ήθελα να θίξω. Καταρχήν θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε την έννοια της ανταγωνιστικότητας. Η ανταγωνιστικότητα δεν γίνεται ευρέως κατανοητή κατά τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη κατανόηση της έννοιας αυτή. Θα πρέπει να εντάξουμε στο κοινωνικό πλαίσιο, όχι μόνο στο χρηματοοικονομικό. Δεύτερον, θα πρέπει να αποφύγουμε αποφύγουμε τις ρήξεις των λόμπι. Διότι ορισμένα αυτά τα, από αυτά τα μέτρα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια σύγχυση και ρήξη σε επίπεδο λόμπι. Θα μπορούσαμε να δούμε πώς έκλεισαν τα ανθρακοριχεία τη δεκαετία του 90 ε, επηρεάστηκαν από τα λόμπι φυσικού αερίου και πετρελαίου και ε, υπό, την συνθήκη ότι δήθεν δεν είναι αποδοτικά αυτά τα ανθρακοειρηχεία, έκλεισαν. Και βεβαίως αυτό οδήγησε σε μεγάλη καταστροφή διότι οι περιφέρειες δεν μπόρεσαν να βρουν εναλλακτικές. Ε, υπήρχαν δυσμενείς ε, κλιματικές συνθήκες και η ανεργία ανέβηκε δραματικά. Τρίτον, τι θα συμβεί εάν εφαρμοστεί αυτό το κριτήριο ανταγωνιστικότητας στις ανανεώσιμες, διότι όλες οι ανανεώσιμες δεν θα ήταν ανταγωνιστικές υπό τους όρους αυτούς. Άρα θα είχαμε ε, δύο μέτρα και σταθμά. Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι ορισμένες ανανεώσιμες έχουν σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. I, I, would say that uh, the first point uh, to start... Όπως στην περίπτωση του ηλαρητικού αερίου. Θα πρέπει να ορίσουμε λοιπόν την έννοια της ανταγωνιστικότητας θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα των ανθρακοριχείων υπό την έννοια των, ε, των, του ανθρώπινου, των ανθρώπινων όρων ζωής και επιβίωσης. Ευχαριστώ. Για να μην ξανακάνω το ίδιο λάθος, θα δώσω τώρα το λόγο στην Κομισιόν. Υποθέτω, κυρία Λεμάν. Ε, καλά τα λέω. Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, θα απαντήσω απλώς σε μερικές ερωτήσεις οι οποίες τέθησαν όσον αφορά ε, τον κανονισμό για το ανθρακά προέβλεπε ότι εκπνέει εφέτος οπότε δεν ε, πρόκειται για προσωπική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά για ένα κείμενο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2011 άρα ένα νέο κείμενο που αναφέρεται στις ε, κρατικές ενισχύσεις. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει ο τομέας αυτός και γι' αυτό έχουμε διατυπώσει προτάσεις για να καλύψουμε την περαιτέρω περίοδο μέχρι το 2010. Ε, μάλλον την ε, περίοδο μετά το 2010. Η, η ε, μελέτη επιπτώσεων έχει γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σύμφωνα με τη γνώμη των ενδιαφερομένων που ελήφθη η υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε σε μια συμβιβαστική λύση προθεσμιών λαμβάνοντας υπόψη και τις κοινωνικές πτυχές και τις περιβαλλοντολογικές που είναι και οι δύο πολύ σημαντικές στον τομέα αυτό. Επίσης οι ενισχύσεις που δίδονται για τον άνθρακα δεν ε, δίνονται σε άλλες ανανεώσιμες πηγές ενεργείας και κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μία στρέβλωση και ε, πρέπει, δεν πρέπει να ε, προωθείται ε, ο τομέας αυτός και γι' αυτό ο, και οι κρατικές ενισχύσεις για την πάση λειτουργία των μπορεί να δοθεί μόνο για μια συγκεκριμένη περίοδο και να μειώνεται συνεχώς. έχετε ερωτήσεις, ναι. Είπατε, είπατε ότι υπήρξαν έρευνες αλλά νομίζω ότι είχατε αναφέρει σαν ημερομηνία ε, την ε, περίοδο μέχρι το 2018. Ε, θα ήθελα να είμαι βέβαιος. σε την αξιολόγηση των ε, επιπτώσεων νομίζω ότι η προθεσμία ήταν μέχρι το 2018 και η υποβολή ε, ε, εκτάκτων κρατικών ενισχύσεων μέχρι το 2026. Κύριε Ζαντό, έχετε τώρα το τελευταίο σχόλιο. Επειδή ετέθη επανειλημμένο ένα ερώτημα, θα ήθελα να ρωτήσω ο κανονισμός μπορεί να αναφερθεί σε επενδυτικές ενισχύσεις γιατί νομίζω ότι αυτό απασχολεί τις, τα μέλη της Επιτροπής δηλαδή θα ήθελαν να μετατρέψουν τις κρατικές ενισχύσεις σε επενδυτικές ενισχύσεις μπορείτε να μας πείτε σε τι αναφέρεται ακριβώς αυτός ο κανονισμός αναφέρεται εις ενισχύσεις για την παραγωγή ε, των μη ανταγωνιστικών ε, ανθρακοριχείων που πρέπει να κλείσουν μέχρι την 1η Ενάτου 2014 των ενισχύσεων που θα συνοδεύσουν ε, το κλείσιμο και μετά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι το 2026 έχετε τον κατάλογο των δυνατοτήτων ε, ε, ως παράρτημα στην πρόταση και μπορεί να ε, ισοσκελίσει το κοινωνικό και το περιβαλλοντολογικό κόστος και εν αντιθέσει προς τον τωρινό κανονισμό δεν προβλέπεται ενίσχυση επενδυτική όπως υπήρχε στον τωρινό κανονισμό για να, ε, για να αναζητηθούν αποθέματα άνθρακα. Ήταν ε, δηλαδή ε, ένα κατάλοιπο του τωρινού κανονισμού που δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ από τα κράτη. Ευχαριστώ κύριε Ζαμπό. Μια τελευταία φορά. Απλώς να πω ότι άκουσα με μεγάλη προσοχή τα σχόλια των συναδέλφων με αυτή την ανησυχία ότι δεν θα αντικαταστήσουμε τα ανθρακοριχεία με εισαγωγές. Δηλαδή τη στιγμή που δίνονται ενισχύσεις για το κλείσιμο ανθρακοριχείων, τότε τα κράτη δεσμεύονται να μην αντικαταστήσουν αυτή τη διαδικασία. Και δεν θα πρέπει να αφήσουμε ολόκληρες ε, περιφέρειες. Εγώ προέρχομαι από μια περιφέρεια που είναι μια ε, ενδυνάμει βιομηχανική έρημος. Δηλαδή θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι χάνονται θέσεις εργασίας, ότι κλείνουν επιχειρήσεις και δεν θα πρέπει να ε, χάσουμε αυτό, αυτό το δυναμικό δημοσίου χρήματος για να κρατήσουμε στη ζωή έναν τομέα ο οποίος πνέει τα λίστια και να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα για άλλες χρηματοκοινωνικές προοπτικές στις περιφέρειες αυτές. Σας ευχαριστώ ειδικά τους συναδέλφους που έμειναν μέχρι τώρα και σας εύχομαι καλό βράδυ. Α, προθεσμία για τροπολογίες. Πέμπτη, 12 η ώρα στα αγγλικά μόνο. Ευχαριστώ, γεια σας.